Αγαπητέ Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλό σας απόγευμα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον πρόεδρο κύριο Ντράγκη για τον ε, διαθρωμένο νομισματικό διάλογο που έχει και ε, ένα ειδικότερο χαρακτήρα σήμερα για δύο λόγους. Πρώτος, διότι Εορτάσαμε πρόσφατα την 20 ετία του ευρώ και στην Ολομέλεια και τώρα είναι η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών αμέσως μετά. Είναι η ιδιαίτερη συνεδρίαση και για έναν άλλο λόγο πρόκειται για την τελευταία εμφάνιση του Πρόεδρου Ντράγκη στην παρούσα Επιτροπή, τουλάχιστον στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αποφασίσαμε λοιπόν να σας προσφέρουμε ένα δώρο κύριε Πρόεδρε για να σας ευχαριστήσουμε για την συνεργασία, την πολύ στενή συνεργασία με την παρούσα Επιτροπή και για το υψηλό επίπεδο διαφάνειας για την κοινοβουλευτική εποπτεία επί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις οποίες υπερασπιστήκαμε και την ανεξαρτησία. Έχουμε λοιπόν εδώ τον νομισματικό διάλογο και τις άλλες μορφές συνεργασίες που έδειξαν ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισχυρή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ταυτόχρονα μιας διαφανούς Κεντρικής Τράπεζας σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλησαμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για αυτό και βέβαια για το συνολικό έργο σας, για όλες σας τις προσπάθειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, για το νόμισμά μας, του οποίου τα 20 χρόνια εορτάσαμε πρόσφατα και πολλοί από τους συναδέλφους μας αναγνώρισαν, και το πράττω και εγώ τώρα, ότι τα όσα πράξατε υπήρξαν θεμελιώδους σημασίας για την διάσωση του νομίσματος, διάσωση του ευρώ, για την προστασία της ακαιρεότητάς του έτσι λοιπόν αποτείουμε φόρο τιμή στις προσπάθειες σας αυτές. Σας ευχαριστούμε και έχουμε όπως ε, σας είπα ένα, ε, μια προσφορά για σας ένα δώρο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Δράγκη. And now, colleagues... Θα θέλαμε να βγάλουμε και μια φωτογραφία με τους ε, υπολείπους συναδέλφους. Αν θέλετε να κατέβουμε κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζει ο πρόεδρος Κουαλτιέρη. Να περάσουμε τώρα στο αντικείμενο του νομισματικού διαλόγου. Ήδη είπα πολλά λόγια. Δεν χρειάζεται να προσθέσω άλλα. Ιδίω άλλωστε διότι έχουμε αναγνώσει όλοι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αξιολόγηση των οικονομικών προοπτικών και την οικονομική πολιτική που παραμένει και τον ευρύ βαθμό ε, των νομισματικών διευκολύνσεων. Σας δίνω το λόγο κύριε Πρόεδρε για να κάνετε τις αγωγικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ευρωβουλευτές της ε, οικονομικής και νομισματικής ε, πολιτικής. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει κάπως από αυτό, πώς να το πω, το δίσκο το δώρο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν έκπληξη για μένα. Κυρίε και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά ξαναβρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον τη δική σα Κοινοβουλευτική Επιτροπή και χαίρομαι που επιλέξατε το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα και τα επιτεύγματα του, τα επιτεύγματα του ευρώ για να συζητήσουμε σήμερα. Θα αρχίσουμε με την ουσία, χωρί άλλη καθυστέρηση θα μιλήσουμε για την εσωτερική και εξωτερική διάσταση του ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι χτίζουμε στα είδη και εκτιμένα, οπότε σήμερα οφείλουμε να συνεχίσουμε την πρόοδο και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα ωφέλη από το ευρώ υλοποιούνται πλήρως. Το ευρώ εισήχθη για να εμβαθύνουμε περισσότερο στην ενιαία αγορά και να διατηρηθεί η καιρότητά της. Συνεχίζουμε λοιπόν το σχέδιό μας για να μειώσουμε τους φραγμούς μεταξύ χωρών και να έχουμε κοινέ πολιτικές. Ακολουθούμε λοιπόν το πνεύμα το οποίο ήδη υπήρχε στη δήλωση του Σούμαν το 1950. Η οικοδόμηση της Ευρώπης δηλαδή μέσω από συγκεκριμένα επιτεύγματα και ως αποτέλεσμα οι οικονομίες μας τώρα είναι ολοκληρωμένες σε βαθμό που κανείς δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί πριν από λίγο καιρό. Το ευρώ σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα σταθερό νόμισμα και αξιόπιστο και όντως καταφέραμε να προσφέρουμε δύο δεκαετίες σταθερότητα στις τιμές. Είχαμε την εμπιστοσύνη του κόσμου όσον αφορά τις αποταμιεύσεις του ευρώ. Επίσης, η σταθερότητα των τιμών διευκόλυναν και τις επενδύσεις, όπως επίσης και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σήμερα έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια παραπάνω Ευρωπαίους στην απασχόληση από ό,τι είχαμε πριν από 20 χρόνια. Στις ε, χώρες δηλαδή που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμα. Και συγχρόνως η συμμετοχή της ε, απασχόλησης, της αγοράς δηλαδή απασχόλησης, έχει ενισχυθεί από το 59% στο 67%. Στις δύο δεκαετίες που έχει υπάρξει το ευρώ, είχαμε πολλές επιτυχίες. Η πρώτη δεκαετία είχαμε 10 ε, χρόνια οικονομικής σταθερότητας, που ήταν γνωστή και ως, ε, ως την μεγάλη επιτυχία αυτού του, της σταθερότητας των τιμών και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φρόντισε να προσαρμόζεται επιτόκια. Στη δεύτερη δεκαετία είχαμε βέβαια την χειρότερη οικονομική κρίση μετά από την μεγάλη ύφεση και είχα την ευκαιρία να συζητήσω βέβαια επί μακρό και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από δύο εβδομάδες ότι ως απάντηση στην κρίση αυτή χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής και να υπάρχει σταθερότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Χάρη λοιπόν στις συλλογικέ προσπάθειες όλων των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωζώνη αναδύθηκε από την κρίση. Τα αποτελέσματα είναι απτά και απο φασιστικότητα όλων μας επίσης ήταν κάτι απτό. Είχαμε ανάπτυξη, είχαμε ε, απασχόληση που σήμερα είναι χαμηλότερη από ποτέ πριν από τον Οκτώβριο του 2008. Όμως, τους τελευταίους μήνες οι εισερχόμενες πληροφορίες συνεχίζουν να είναι από ό,τι αναμενόταν λόγω της υπιότερης εξωτερικής ζήτησης σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένους τομείς. Έτσι παραμένει αβεβαιότητα κυρίως λόγω γεωπολιτικών παραγόντων και η απειλή επίσης του προστατευτισμού επηρεάζει την κατάσταση. Συγχρόνως, οι υποστηρικτικέ συνθήκε χρηματοδότηση, η ευνοϊκή δυναμική των αγορών εργασία και η επιταχυνόμενη άνοδο των μισθών συνεχίζουν να στηρίζουν την επέκταση τη ζώνη του ευρώ και τις σταδιακά αυξανόμενες πιέσεις στον πληθωρισμό. Αυτό στηρίζει την πεποίθησή μας ότι θα συνεχιστεί η διαρκή σύγκληση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίων του 2% μεσοπρόθεσμα. Επίσης, η νομισματική, σημαντική, η νομισματική μας πολιτική είναι βασική για να στηριχθούν οι παρετέρω συσσόρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές και οι εξελίξεις στον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Αυτό θα γίνει με τις ενδείξεις μας για την μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες θα ενισχύονται από τις επανεπενδύσεις του σημαντικού αποθέματος αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει αναλόγως όλα τα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται διαρκώς προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξη του Δικητικού Συμβουλίου για τον Πληθωρισμό. Το ωφέλη από, από το ευρώ δεν περιορίζονται βέβαια στην εσωτερική ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί μαζί, στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, μπορέσαμε να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας, η οποία θα είχε χαθεί από επιμέρους χώρες μέσα σε, έναν, σε μια οικονομία παγκοσμιοποιημένη. Κάτι το οποίο το ξέραμε ήδη από τη δημιουργία του ευρώ. Συμβολίζει το ευρώ την ενότητα της Ευρωπαϊκής Υπήρου που έτσι μπορεί καλύτερα να επηρεάσει διεθνώς τα πράγματα. Το ότι είμαστε μαζί στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μας ε, επιτρέπει να έχουμε πιο δυνατή φωνή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και ενισχύει επίσης την ικανότητά μας να επηρεάζουμε τις οικονομικές σχέσεις. Αυτά τα είπε ο Ζακ Ντελόρ στην περίφημη έκθεση Ντελόρ. Τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν το ευρώ έγινε το δεύτερο πιο σημαντικό νόμισμα στο διεθνές νομισματικό σύστημα κάπου ανάμεσα στο 20 και 40% του αποθεματικού και των συναλλαγών διεθνώς, όπως επίσης και στο χρέος και σε άλλες συναλλαγές, είναι σε ευρώ. Και πάνω από 50 χώρες οι επικράτειες χρησιμοποιούν ή συνδέουν το νόμισμά τους με το ευρώ. Αυτή η παγκόσμια κατάσταση αποφέρει ωφέλη γιατί μειώνει το κόστος συναλλαγών στις διεθνείς συναλλαγές και η Ευρωζώνη έτσι γίνεται πιο ανταγωνιστική. Επίσης, προσθέτει και ρευστότητα στην ε, αγορά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επιτρέπει έτσι στους επενδυτές στο εσωτερικό αλλά και απ' έξω να μπορούν να υποφεληθούν και να δώσουν πόρους με μεγαλύτερη άνεση. Επίσης για τους δανειστές, για τις εταιρείες, για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν εμπιστοσύνη τα νοικοκυριά, οι φορολογούμενοι. Βέβαια, ο διεθνής ρόλος του ευρώ φέρνει μαζί και προκλήσεις. Εκτίθεται περισσότερο στις ε, εξελίξεις παγκοσμίω και στις αλλαγές στην ε, νομισματική πολιτική τα διεθνή ωφέλη του να έχουμε ένα κοινό νόμισμα ξεπερνούν το νομισματικό σκέλος. Μέσα σε ένα κόσμο όπου συνδέονται τα οικονομικά, σε κάθε επίπεδο η διεθνή συνεργασία είναι ζωτική σημασία και μπορούμε πιο αποτελεσματικά να προωθήσουμε τι ευρωπαϊκέ ιδέε και τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά εφόσον μιλούμε με μία φωνή. Η φωνή της Ευρωζώνης ήταν ζωτική σημασία και μπόρεσε να ενισχύσει το δημοσιονομικό ρυθμιστικό πλαίσιο μετά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Σήμερα, ο ενιαίος εποπτικός ο μηχανισμός είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός εποπτικός μηχανισμός παγκοσμίω και διαμορφώνει το διεθνές ε, ρυθμιστικό εποπτικό σύστημα. Μετά την ε, κρίση ε, χρέους στην Ευρωζώνη και αλλού, ο διεθνής ρόλος του ευρώ φάνηκε να διαβρώνεται. Και ενώ είναι πολύ σημαντικό στις διεθνείς συναλλαγές το ευρώ, ο ρόλος του παρέμεινε σταθερός. Στα αποθεματικά διεθνώς έχει μειωθεί. Αυτή η μείωση αποτελεί ένα σύμπτωμα της έκθεσης λόγω της κρίσης ανησυχίες για την αντοχή του ευρώ και της οικονομικής και νομισματικής αρχιτεκτονικής του ευρώ, ο κατακαιρματισμός υπογραμμίζουν ακριβώς αυτήν την διαβροτική τάση. Η σταθερότητα, η ρευστότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες για ένα διεθνές νόμισμα. Εκείνοι που καταρτούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές τα έχουν διαπιστώσει όλα αυτά όλους αυτούς τους μήνες και φροντίζουν προκειμένου το ευρώ να μπορεί να παίξει έναν περισσότερο ισχυρό ρόλο διεθνώς. Η διάσκεψη του Δεκεμβρίου του 2018 μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε τη δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο διεθνής ρόλος του ευρώ στηρίζεται από από υγιείς νομισματικές πολιτικές στην Ευρωζώνη και από την ευάθυνση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό απαιτεί περισσότερες προσπάθειες για περισσότερη ακόμα ολοκλήρωση. Τα τελευταία 20 χρόνια, δίχως άλλο, έδειξαν πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσουμε, τη, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι μάλλον η σταθερότητα και η ευημερία οικονομική. Και αυτό φάνηκε τόσο μέσα στην Ευρωζώνη αλλά και εκτός αυτής. Παρόλα αυτά, Όλα αυτά τα χρόνια μας έδειξαν ότι αυτή η επιμερισμένη πρόκληση αντιμετωπίζεται καλύτερα όταν την αντιμετωπίζουμε μαζί. Όταν διαπιστώσουμε ποια είναι τα ωφέλη από το ευρώ, πρέπει να έχουμε τα ίδια συστατικά όπως είχαμε και πριν από το ευρώ. Χρειαζόμαστε όμως συγχρόνως και μεταρρυθμίσεις για να έχουμε περισσότερη ανθεκτικότητα. Υπάρχει αναπτυξιακό δυναμικό, το οποίο όμως θα επιτευχθεί μόνο εφόσον συνεχιστούν οι προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά τώρα την σύγκληση, που εξαρτάται βέβαια και από διορθωτικούς παράγοντες, αυτό είναι ευθύνη των χωρών μελών. Από την άλλη, η Ευρώπη μπορεί να κάνει τη διαφορά, στηρίζοντας και διευκολύνοντας τέτοιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στις χώρες μέλη το να είμαστε μαζί αποτελεί ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μας και πρέπει να αποφεληθούμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να χτίσουμε στις ε, συνέργειες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας αγοράς. Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να απελευθερώσουμε τους μηχανισμούς ε, οι οποίοι θα βοηθήσουμε τη σειρά τους στην ε, παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στην χρηματοδότηση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Χρειάζεται καινοτομία και όλα αυτά μπορούμε να τα, μετύχου, τα πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται επίσης διαφοροποίηση που θα διευκολύνει την περίπτωση κάποιας ύφεση σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Έπειτα είναι πολύ βασικό να ολοκληρωθούν τα σχέδια τα οποία ξεκινήσαμε ε, με την κρίση, την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιογορών. Μια ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση θα μας βοηθήσει για περισσότερα ωφέλη ακόμα, κάτι το οποίο δεν έχουμε σήμερα να το συγκρίνουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να υπάρχει στήριξη και από άλλες πολιτικές. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να το καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό υπέρ οικονομιών που να είναι στέρεες και ανθεκτικές. Υπάρχει απόφαση πρόσφατα να ξεκινήσουμε ένα μέσον για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα για την ε, Ευρωζώνη. Προκειμένου να πετύχουμε επίση την αντιμετώπιση μελλοντικών ε, κυκλικών ε, κρίσεων, χρειάζεται διαφοροποίηση του κινδύνου μέσα από το ιδιωτικό σύστημα χρηματοδότησης αφενός και μέσω αντικυκλικής στήριξης από το δημόσιο με μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούμε έτσι να είμαστε αποτελεσματικοί για να πετύχουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, μάλλον δεν λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις ε, έτσι απλώς σαν όνειρο ή ότι είναι τοπικό, όχι, αν συνεργαστούμε και είμαστε μαζί θα το καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν το Δεκέμβριο οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αν θέλουμε να αποφεληθούμε πλήρως από το ωφέλη του ευρώ, πρέπει να κεφαλοποιήσουμε ακριβώς πάνω σε αυτή τη δέσμευση και να την ε, καταστήσουμε πραγματικές δράσεις για την οικονομία μας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλές φορές είπα μαζί σήμερα. Μίλησα για αυτό το μαζί και επειδή είναι η τελευταία φορά που θα είμαστε μαζί εδώ, σε αυτήν τη θητεία, επιτρέψε μου για σας προσωπικά να προσθέσω κάποια λόγια. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τον ρόλο της δικιάς σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη μου ακρόαση εδώ θυμάμαι ότι είπα πως ήταν η πρώτη άσκηση που έκανα όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπα ότι ήμουν πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία αυτή. Πολλές τέτοιες ακροάσεις ακολούθησαν και διασφαλίσατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πράγματι λογοδοτεί και παραμένει ανεξάρτητη όταν φέρνει σε πέρας την οικονομική γνωμοσματική πολιτική. Αλλά θέλω επίση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξη τη δικιά σα επιτροπή στι δικέ μα προσπάθειε. Ήταν ουσιαστική γιατί χτίζεται πάνω στην φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και είναι μια στήριξη που βοήθησε πολλές φορές τους δύσκολους καιρούς που περάσαμε τελευταία την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως νομοθέτες, ο δικός σας ρόλος ήταν ουσιώδης για να πετύχουμε βασικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ένωσή μας. Η Επιτροπή αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την εμπειρία που έχω εγώ, βοήθησε ουσιαστικά να πάμε πιο κοντά στον πολίτη και μόνο έτσι υπάρχει εμπιστοσύνη για την νομιμότητα των θεσμών και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι εφικτό να πετύχουμε μια πιο αποτελεσματική ένωση με τη συμμετοχή όλων. Οι πολίτες ζητούν και μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πετύχουμε μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη, η οποία να συνεχίζει να προσφέρει στους πολίτες και φυσική αλλά και οικονομική προστασία και στήριξη μέσα σε μια δημοκρατική και ειρηνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για, τη, για τα ευγενικά σας λόγια σχετικά με τις δραστηριότητες της παρούσης Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Ας αρχίσουμε τώρα με τις παρεμβάσεις των μελών μας και πρώτον τον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Συγγνώμη που θα σας μιλήσω γερμανικά, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να τα καταφέρω να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα, ως βαβαρός εννοώ Ευχαριστώ στο όνομα της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε, για τον πάντα ανοιχτό τρόπο με τον οποίο ε, προσεγγίσατε τον... Ε, επαναλαμβάνω. Ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα λοιπόν στο όνομα της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον πάντοτε ανοιχτό τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε τον οικονομικό διάλογο και για τις πολλές δυνατότητες που μας δώσατε να συνομιλήσουμε όχι μόνο στην ε, Επιτροπή μας αλλά και συχνά στην Φραγκφούρτη αλλά και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπήρχε δυνατότητα δηλαδή να συναντηθούμε. Αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερος και έχετε βάλει και τον πύχη αρκετά υψηλά για τους διαδόχους σας. Επιτρέψτε μου δύο ερωτήσεις. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διαγράφει πώς βλέπει τον διεθνή ρόλο του ευρώ και ιδίως τον ρόλο του ως αποθεματικού νομίσματος. Ποιες είναι οι επιπτώσεις που προκύπτουν για σας από αυτό το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, χρηματική πολιτική, για την νομισματική πολιτική και θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μάλλον, παίζει μια πιο περιοριστική ε, εξασκεί μια πιο περιοριστική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει την νομιμότητα των εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο προπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επομένω και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ακούσαμε για την εποπτεία του εποπτικού μηχανισμού. Ξαναλέω λοιπόν, συνολικός εποπτικός μηχανισμός και δυνατότητα αντίδραση σε, κρίσεων, σε κρίσεις. Ακούσαμε λοιπόν κατ' επανάληψη την δήλωση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν διαθέτει, δεν δίνει δηλαδή σε επαρκή βαθμό τα αναγκαία έγγραφα για να μπορέσει το ελληνικό συνέδριο να ασκήσει τον έλεγχο. Μπορείτε να εξηγήσετε για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρεί σε επαρκή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τι προτίθεται να κάνετε για να βελτιωθεί αυτό. Πρόεδρος Δράγκη, δύο ερωτήσει μου κάνατε. Πρώτα, πώς θα επεκταθεί, ο, μάλλον πώς ο εκτεταμένος διεθνής ρόλος του ευρώ επηρεάζει την νομισματική πολιτική. Πρέπει να ρωτήσουμε πρώτα γιατί ο διεθνής μας ρόλος δεν είναι τόσο μεγάλος όσο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς λόγω του μεγέθους της Ευρωζώνης. Και η απάντηση είναι βασικά απλή. Ολοκληρώστε την Τραπεζική Ένωση και από τη στιγμή εκείνη και μετά θα έχουμε έναν διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα που θα είναι ανάλογος με αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος του ευρώ θα είναι το ίδιο μεγάλος και κυρίαρχος όπως του Αμερικανικού δολαρίου. Τώρα, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι δεσμοί μεταξύ του ρόλου της Ένωσης και της νομισματικής πολιτικής, αλλά βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη όσα κάνουμε τώρα και τα spillover από και προς άλλες δικαιοδοσίες. Λαμβάνουμε υπόψη τα spillover σήμερα, αλλά ο σύνδεσμος θα γίνει αμεσότερος σε ένα τέτοιο μέλλον. Σε ό,τι αφορά μια χαλαρή νομισματική πολιτική. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε άρχισαν την ποσοτική χαλάρωση μερικά χρόνια πριν από εμάς και τώρα σταμάτησαν. Αλλά είναι και σε τελείως διαφορετική θέση στον επιχειρηματικό κύκλο, στο business cycle. Δεν συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με την χαλαρότητα της νομισματικής πολιτικής. Αλλά, ξαναλέω, οι Ηνωμένε Πολιτείε άρχισαν πολύ πριν από εμά για την πρώτη σας ερώτηση αυτά. Για τη δεύτερη ερώτηση, για το ελεγκτικό συνέδριο. Θα μπούμε και σε λεπτομέρειες, αλλά κατά βάση εμείς συνεργαζόμαστε. Έχουμε παραγάγει 500 έγγραφα μετά από αίτηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Συνολικά 6.000 σελίδες, 38 συναντήσεις και διασκέψεις με το ελεγκτικό συνέδριο. Και τους παρέσχομαι όλες τις προφορίες που ζήτησαν εντός των αρμοδιοτήτων, των πλαισίων αρμοδιοτήτων των δύο θεσμικών οργάνων. Η συνθήκη δηλώνει ότι το ελεγκτικό συνέδριο καλείται να ε, εξετάσει και να ελέγξει την αποτελεσματικότητα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά λέει ο νομοθέτης για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 συμφώνησε με την νομική ερμηνεία που κάνουμε εμείς του καταστατικού μας. Τούτου λεχθέντος, όπως είπα και πριν, έχουμε συνεργαστεί ευρύτατα. Αλλά, ξαναλέω, μέσα στα πλαίσια της εντολής μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μπερές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος Σώματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κεντρικής Τράπεζας στη διάρκεια της ε, θητείας σας. Η κατάσταση εξελίχθηκε. Θα το θυμάστε ασφαλώ ότι η πρώτη ακρόαση, όταν ήσταν ακόμη υποψήφιος, διοικητή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σας είχα εγώ απευθύνει σε εκείνη την ακρόαση μια αρκετά σκληρή ε, ερώτηση και θέσεις. Κάποιοι φίλοι που είχαν καλή γνώση των οργάνων μου είχαν πει ότι ε, θα ε, μπορούσατε να αποδειχθείτε σπουδαίος διοικητής Κεντρικής Τράπεζας λόγω των γνώσεών σας. Και όντως το πράξατε αυτό, σας συγχαίρω. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω καταρχάς πώς εκτιμάτε την κατάσταση ως προς τις συνέπειες των δημοσιονομικών πολιτικών. Γιατί έχουμε την εντύπωση πως ε, η πολιτική που εφαρμόζεται έχει να κάνει ιδιαίτερως με την υποτίμηση των δημοσιονομικών πολιτικών. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Δεύτερον, για να συνεχίσω στα όσα είπε ο κύριος Φέρμπερ. Ε, γιατί έχω την εντύπωση πως ε, η αναζωγόνηση αυτής της συζήτησης για την ε, παγκόσμια κτηνοβολία του ευρώ μπορεί να θεωρείται και λίγο σαν διέξοδος, αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ακριβώς το γεγονός ότι δεν είναι ολοκληρωμένο το ευρώ και δεν έχει το σύστημα το, της διαχείρισης και το χρηματοπιστωτικό ε, είναι εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο για το ότι δεν έχει την ακτινοβολία σε παγκόσμιο σκηνικό. Αλλά τι νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να πούμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο στην κατεύθυνση αυτή. Απάντηση. Για την πρώτη σας ερώτηση. Αυτό που πρέπει να αποφεύγει παντού βέβαια, αλλά και κυρίως στη δική μας την περίπτωση μια νομισματική πολιτική, είναι η δημοσιονομική επικράτηση. Η δάλος χάνει την ανεξαρτησία της και άρα και την αξιοπιστία της η Κεντρική Τράπεζα. Υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν, όχι στην Ευρωζώνη, αλλά σε άλλες περιοχές του κόσμου ή θα έλεγα πριν από το ευρώ ακόμη, πριν από την εισαγωγή του ευρώ, όπου κεντρικές τράπεζες επηρεάζονταν σημαντικά από τα δημοσιονομικά μελήματα και θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι έχασαν κατά κάποιο τρόπο την ανεξαρτησία τους και άρα σε συνέπεια αντιμετώπισαν και ποσοστά ε, πληθωρισμού και ποσοστά ανεργίας πολύ υψηλά. Αυτό το είδαμε στη δεκαετία του 80 κυρίως. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο που θα πρέπει να κοιτάξουμε τώρα του Τουλεχθέντο. Μπορούμε να βελτιώσουμε τους υφιστάμενους δημοσιονομικού κανόνες. Ή να γυρίσω λίγο πίσω. Μεγάλη διαφορά βλέπω μεταξύ της δημοσιονομικής και της νομισματική πολιτικής ως προς την ολοκλήρωση. Στον χώρο της οικονομικής πολιτικής από τη δεκαετία του 80 όπου η ενοποίηση και ο συντονισμός των πολιτικών εξασφαλίζονταν από κανόνες ένα σύστημα δηλαδή στηριζόμενο σε κανόνες και όπου καταγράφηκε στη συνέχεια η αποτυχία του συστήματος αυτού και έτσι οι ιδρυτές του ευρώ πέρασαν σε μια θεσμική ενοποίηση των νομισματικών μας πολιτικών. Αυτό προέκυψε ύστερα από 15-20 χρόνια αποτυχιών του συστήματος που στηριζόταν σε κανόνες. Στη δημοσιονομική πολιτική όμως αυτό δεν έχει ακόμα ε, υλοποιηθεί γιατί ακόμη ακολουθούμε κανόνες, το σύστημα των κανόνων. Και έτσι μπορεί τώρα βέβαια να είναι του σειρμού να επικρίνονται αυτοί οι κανόνες. Ωστόσο θεωρώ πως απεδείχθησαν πολύ χρήσιμοι. αν διανοηθούμε παραδείγματι πώς θα είχαν τα ελλείμματα και τα χρέη εξελιχθεί εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι κανόνες. Βεβαίως, οι κανόνες και βεβαίω μπορούν να βελτιωθούν οι κανόνες και πρέπει να βελτιωθούν. Στους επόμενους μήνε τα επόμενα χρόνια πρέπει να εξασφαλίσουμε βελτίωσή τους. Εν τέλει όμως, και το έχω πει και με άλλη ευκαιρία, ο καλύτερος συντονισμό θα πρέπει να στηρίζεται και σε θεσμούς, όπω στην νομισματική πολιτική. Για το διεθνή ρόλο του ευρώ. και νομίζω ότι είναι εύστοχη η πρόκληση αυτή τη συζήτηση γιατί μας αναγκάζει να κοιτάξουμε τι συμβαίνει εκεί όπου τα νομίσματα έχουν πολύ μεγάλο διεθνή, πολύ μεγάλη διεθνή αντανάκλαση όπως το αμερικανικό δολάριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και έχουμε μια καλά λειτουργούσα κεφαλαιοχική αγορά, κεφαλαιακή αγορά και τραπεζική ένωση με έναν έχουν συγγνώμη, με έναν προπολογισμό και μια κυβέρνηση. Και εμεί δεν είμαστε μία χώρα, αλλά πολλέ χώρε. Και άρα πρέπει να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση εκείνη που θα μα επιτρέψει τον μεσματικό μα χώρο να τον, να τον βελτιώσουμε, γιατί ακόμη δεν έχει φτάσει στο ιδεούδε. Έχει πολλά σημεία ευάλωτα, άλλωστε το διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και ταυτόχρονα σταδιακά και με τις πολιτικές εξελίξεις διάφορες χώρες προχωρούμε προς την κατεύθυνση αυτής της ενοποίησης. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Τράγκη, σας ευχαριστώ επίσης για τα φιλικά λόγια που απευθύνατε προς την Επιτροπή μας, έστω και εάν οφείλω να ομολογήσω ότι δεν συγκαταλέγω μεταξύ εκείνων που θα συνεργαστώ μαζί σας ε, για την ολοκλήρωση της υπόθεσης του ευρώ, γιατί εξακολουθώ να θεωρώ ότι το ευρώ δεν είναι κατάλληλο νόμισμα για την Ευρωζώνη ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και γιατί δεν συμφωνώ με την αντίληψή σας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τηρεί όντω την εντολή της. Εγώ θεωρώ ότι την υπερβαίνει, όπως άλλωστε το γνωρίζετε. Κατά τούτο, λοιπόν, βρισκόμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα. Ομολογώ ότι είστε καλός ε, μαχητής, αν θέλετε, αλλά για τη λάθος αιτία. Σας ευχαριστώ βεβαίω για τον τρόπο με τον οποίο έχετε διεξαγάγει ως τώρα τον ε, νομισματικό διάλογο έως τώρα και που πραγματικά ε, είναι από τους καλύτερους τρόπους που έχω ζήσει ποτέ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα επιχείρηματά σας η διάρθρωση των επιχειρημάτων σας όλα είναι πραγματικά υποδειγματικά και σας ευχαριστώ πραγματικά διότι επιτρέψατε ένα αληθινό διάλογο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το θόλωμα αυτό της ε, διαρθρωτικής κατάστασης όπως εμφανίζεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι το PSPP έχει μειωθεί τώρα και δεν πρόκειται να γίνουν νέες καθαρές αγορές. Εν όψη όμως του γεγονότος ότι το PSPP εξακολουθεί να παραμένει στην φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, θεωρείται ενδεχόμενο οι καθαρές αγορές μέσα στα πλαίσια του 2019 επαναληφθούν για να, δοθεί, να δοθούν εκ νέου κίνητρα και όθηση στην οικονομία και ποιοι λόγοι ενδέχεται να το καταστήσουν αυτό αναγκαίο κατά την άποψή σας. Η δεύτερη ερώτηση, ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά μαζί για τους στόχους. Δηλαδή θα έχετε μάθει ότι υπάρχει μελέτη των καθηγητών Φούστ και Ζιν, οι οποίοι προβάλλουν το επιχείρημα ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στην εσωτερική σχέση του συστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορούν να είναι αφαιρέγγιες, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε φυγή κεφαλαίων, όπου οι υποχρεώσεις πληρωμών που προέρχονται από τα, που θα καταλήξουν δηλαδή στους ολογισμούς παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό που λέω ή ενδεχομένως μπορείτε να αποκλείσετε ότι μια εθνική κεντρική τράπεζα σε ένα τέτοιο σενάριο, σαν αυτά δηλαδή που σχεδιάζουν οι και Ζήν στη μελέτη τους, μέσα στην εσωτερική σχέση των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών μπορεί να, μπορεί να καταστούν αφαιρέγγιες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις ευχαριστίες σας τις οποίες εκτιμώ ακόμη περισσότερο, διότι όπως είπατε προέρχονται από κάποιον ο οποίος πρεσβεύει πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά ε, τα, οποία, ε, τα οποία υπερασπίζομαι εγώ. Αλλά πρώτα θα ήθελα ε, να θίξω ένα θέμα για την εντολή μας, διότι συνδέεται και με το υπόλοιπο της απαντήσεως. Μπορεί κανείς να έχει υποκειμενικές αμφιβολίες για το εάν κάποιες δράσεις εμπίπτουν στην εντολή ή όχι. Το γεγονός όμως είναι ότι το ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκύρωσε το γεγονός, επεκύρωσαν δηλαδή το γεγονός, ότι εμείς δρούμε εντός της εντολής και ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι τμήματα της νόμιμης εργαλειοθήκης μας που χρησιμοποιούμε και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Έρχομαι τώρα μέσα στην ερώτησή σας. Όπως είπα, έχουμε ε, διάφορα εργαλεία, έχουμε τη Forward Guidance για τα επιτόκια, που είναι σχέση, έχει σχέση και με τον χρόνο, με, το, με την ημερομηνία δηλαδή, αλλά και με τις χώρες. Δεν προχωρούμε πλέον σε καθαρή βάση σε αγορές ε, στοιχείων ενεργητικού. Συνεχίζουμε να αγοράζουμε ομόλογα μόνο για να σταθεροποιήσουμε το απόθεμα, όταν φτάνουν σε οριμότητα, σε λήξη δηλαδή τα ομόλογα αυτά. Έχουμε τη forward guidance, έχουμε και τις επανεπενδύσεις των αποθεμάτων ομολόγων που θα είναι και αρκετά μεγάλα τούτη εδώ τη χρονιά διότι μιλούμε για 50 δισεκατομμύρια τον μήνα. Και βέβαια εάν τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα μπορούμε πάντοτε να επανέλθουμε στην χρήση άλλων εργαλείων που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας. Ένα από τα οποία είναι αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία, κανένας είδους ένσταση σε αυτή τη δυνατότητα. Το άλλο ερώτημα είναι υπό ποιους όρους θα το πράξουμε αυτό. Επί του παρόντος δεν βλέπουμε να διαγράφονται τέτοιες περιπτώσεις ως πιθανόν να υλοποιηθούν δηλαδή φέτος και σίγουρα όχι φέτος πάντως. Για το δεύτερο ερώτημα. Ε, ρωτήσατε τι γίνεται εάν. Δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες για ενδεχόμενα που μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Μπορώ να πω λίγα λόγια για την υποκείμενη αυτή ανησυχία που αποκαλύπτει η ερώτησή σας, δηλαδή την αύξηση στις, ε, στους του στόχου 2. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και αλλού, αλλά ο, ο βασικός θεμελιώδης παράγων πριν, πίσω μάλλον από την αύξηση αυτή είναι η αποκέντρωση της εφαρμογής της νομισματικής μας πολιτικής και εξαρτάται κυρίως από την νομισματική μας πολιτική, από το QE, από τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού, εάν θα αυξηθούν αυτές οι πολιτικές στόχου 2. Κάθε φορά δηλαδή που οι πληρωμές κεντρικών τραπεζών ρυθμίζονται διαμεθοριακά, μπορεί να επηρεάσουν τους στόχους, της ε, ισολογισμού στόχου 2. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν αυτούς τους ισολογισμούς από αυτήν την οπτική. παρακολουθούμε τις αυξήσεις που αποκλίνουν από την τάση αυτή. Τις μεγαλύτερες δηλαδή αυξήσεις του στόχου 2. Και πρέπει να τις παρακολουθούμε. Αλλά έχουμε αυξήσεις των ε, ισολογισμών στόχου 2 σε ορισμένες χώρες και αλλού μειώσεις. Είναι λοιπόν δύσκολο λοιπόν να εκτιμήσουμε εάν ακολουθούν εδώ αυτές οι balances κάποια, κάποιες τάσεις. Και πιο γενικά, σε κάθε νομισματική ένωση έχετε, θα έχετε χώρες οι οποίες θα βρίσκονται σε κατάσταση ελλείμματος, άλλες οι οποίες θα βρίσκονται σε κατάσταση πλεονάσματος. Και αν εξετάσουμε και τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι ασφαλώς τελειότερη νομισματική ένωση, έχετε ένα status quo από την αρχή, εδώ και 200 χρόνια, από την αρχή της ύπαρξής τους και η νομισματική ένωσή τους λειτουργεί καλά. Το βασικό εδώ είναι, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε διαφορετικές οπτικές, αλλά το βασικό εδώ είναι, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, όχι τόσο να τεθεί το ερώτημα εάν μπορεί μια χώρα, αν μπορεί μια κεντρική τράπεζα να είναι αφαιρέγγια. Το αντίθετο ερώτημα, Το σύστημα πληρωμών της Νομισματικής Ένωσης λειτουργεί αποτελεσματικά. Και η απάντησή μου είναι ναι. Σας ευχαριστώ. Καρολίν Μακδούγκαλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Πρόεδρε Μπτράκη που είστε εδώ. Έχω δύο ερωτήσει. Η πρώτη έχει να κάνει με τις οικονομικές προβλέψεις που την προηγούμενη εβδομάδα κατέκλυσαν τον νιοσφίτ μου με την πρόβλεψη για μείωση των εμπορικών συναλλαγών. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε πώς προξενούν ε, και οι προστατευτικές τάσεις του Brexit αλλά και οι επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ, Τραμπ και ενδέχεται να επηρεάσουν την παγκόσμια ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να καθισχάσει να μπορείτε το Κοινοβούλιο όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει περιθώριο χειρισμών επαρκές σε περίπτωση σημαντικής οικονομικής επιβράδυνσης. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη και κάπως πιο τεχνική σε σχέση με τα ορόσημα, benchmark. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, εξασφαλίζει τη γραμματική υποστήριξη στην ομάδα εργασίας για τον κόσμο χωρίς κινδύνους Risk Free ε, World Working Group και βλέπω ότι με ικανοποιήσει ότι ε, χορηγεί και τα σχετικά ορόσημα. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν κάποια στοιχεία για τη μετάβαση της Ενωνία και της Έσταρτα Νέα, δηλαδή benchmark που έχει εξασφαλίσει, που έχει ε, καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θεωρείται πως οι ε, μετέχοντες στην αγορά, οι φορείς που προστατεύονται στην αγορά θα τα δεχθούν έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Τελευταία ερώτηση. Η Euribor μετατρέπεται πλέον σε μια πιο υβριδική μορφή σε κάποιο βαθμό εξαρτάται, στα, εξαρτάται από τα πάνελ και δεδομένων των ε, περιθωρίων για συμβολή στο Νιαμάρ θεωρείται ότι μπορεί να είναι ασφαλής η διαπίστωση ότι οι επιλογές γίνονται μόνο με βάση στοιχεία και τεκμήρια. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίστηκε πως η τάση ανάπτυξης αρχίζει να παρουσιάζει μειωτική ε, πορεία με λόγους αυτούς ή κάποιους εκ των λόγων που εντοπίσαμε, αυτούς ε, τους οποίους και εσείς επισημάνατε. Πριν απαντήσω προς την πολιτική. Η συστήση στο Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι ο κύριος παράγων πρέπει να εξετάσουμε είναι η έμονη παρουσία αυτών των διαφόρων, η μόνιμη παρουσία αυτών των διαφόρων παράγοντων, ο προστατευτισμός, παραδείγματι. γιατί ήταν πολλά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είπαν ότι εάν ξαφνικά επικρατήσει ειρήνη στις εμπορικέ συναλλαγέ και σαφήνεια στη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ιδιαίτερω, πολλά από τα προβλήματα αυτά θα ε, εκλείψουν. Ε, άλλη πηγή προβλημάτων είναι οι ανησυχίες ε, που προξενούν οι συνομιλίε και την πραγματεύση για το Brexit. Είπατε κι εσείς ότι ίσως αυτό να μην σημάνει απαραίτητα σε πραγματικούς όρους πρόβλημα και ότι υπάρχουν πολλές, κάποιες χώρες οι οποίες είναι πολύ εκτεθειμένες στις συναλλαγές ε, ή στις συνέπειες του Brexit, αλλά άλλες λιγότερο. Και κάτι ακόμη, η αλυσίδα παραγωγής αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περίπλοκη, άρα δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κάποια ε, ε, κάποιες τοπικά προσδιορισμένες συνέπειες αυτής της δυσφορίας. Ε, το ότι καθυστερούν και μόνο αυτές οι διαπραγματεύσεις τροφοδοτεί την ανησυχία. Και βεβαίως και οι γενικές πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, η επιβράδυνση της οικονομικής ε, δραστηριότητας της Κίνας ε, και τι, πιστεύουμε πως και εκεί η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις, τα κατάλληλα μέτρα. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητική η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση στο πρόβλημα αυτό ή τα προβλήματα που μπορεί να προξενεί η δημοσιονομική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να έχουν πολιτικη στι ΗΠΑ πολιτειες κάποια προβλήματα. Πάντως γενικά ως προς τη χάραξη πολιτικής μπορώ να απαντήσω πως ναι, έχουμε μέσα εργαλεία τα οποία ήδη σε ένα βαθμό έχουν αρχίσει να φέρουν αποτελέσματα χάρη στην ενισχυμένη και προληπτική καθοδήγηση που έχουμε. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως μέχρι το καλοκαίρι και πάντως, ή αν μου επιτρέπετε να αναγνώσω το σχετικό κομμάτι, συνεχίζουμε να περιμένουμε πως ε, ε, τα επιτόκια θα διατηρηθούν τα, της Κεντρικής Τράπεζας θα, παραμένουν, θα διατηρηθούν μέσα στο καλοκαίρι του 2019 και πάντως έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθήκων ρευστότητας και ενός διευκολυντικού σε μεγάλο βαθμό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής. Και για να περάσω στο τομέα που αφορά τις επενδύσεις, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πλήρη βαθμό το πρόγραμμα αγορά στοιχείων ενεργητικού λοιπόν για μια ε, παραταταμένη χρονική περίοδο έχει ήδη ξεπεράσει, έχει συνεχιστεί δηλαδή και μετά την περίοδο κατά την οποία έγινε η αύξηση του επιτοκίου και όσο χρειάζεται για την ε, εξασφάλιση ευνοϊκών ε, συνθήκων ρευστότητας και ενός διευκολυντικού σε μεγάλο βαθμό χαρακτήρα της ομασματικής πολιτικής. Άρα, ο ορίζον των επενδύσεων διαφυλάσσεται στο μέλλον και βλέπουμε ήδη άμεσα αποτελέσματα μετά την ανακοίνωση του τέλους του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού πέρσι τον Ιούνιο που δεν είδαμε αντίδραση των αγορών δυσμενή. Και μάλιστα όταν ακόμα μειώθηκαν τα επιτόκια συμπιέστηκε η δομή τους και μετακινήθηκε όπως λέμε προς τα δεξιά. Δηλαδή τις προβλέψεις για περαιτέρω ε, μειώσει τα επιτόκια, αυξήσει τα επιτόκια τις μεταφέρει σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το καλοκαίρι δηλαδή χρονικά. Αυτό σημαίνει μια πολύ πιο μετριοπαθή αντίδραση στον κίνδυνο της επιβράδυνσης. Άρα λοιπόν όχι μόνο έχουμε στην εργαλειοθήκη μας τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά έχουμε ήδη αρχίσει, έχουν ήδη τα εργαλεία αυτά αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα αντιμετωπίζοντα την επιβράδυνση. Για τα ορόσημα. Benchmark. Είπατε κι εσείς ότι η διοίκηση του Euribor ήδη επεξεργάζεται μια μεταρρύθμιση έτσι ώστε να το ευθυγραμμίσει με τις προϋποθέσεις ε, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα benchmark. Άρα το τελικό, την τελική έκβαση των προσπαθειών αυτών θα την δούμε προς τα τέλη του έτους. Εν τω μεταξύ, η ομάδα εργασίας ε, καταργάσετε ένα σχέδιο με το οποίο ίσως να μην προσαρμόζεται το Euribor στους κανόνες. Βεβαίως δεν θέλουμε να σχολιάσουμε ένα τέτοιο σενάριο, αλλά πάντως οπωσδήποτε πρέπει να αναλυθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεδομένου ότι ο εντοπισμός πιθανών λύσεων είναι, ανήκει στον ιδιωτικό τομέα μαζί με τις εποπτικές αρχές, φύσμα και έσμα δηλαδή, για δε την ε, πιθανή παραγωγή επιτοκίου, περιοδικού επιτοκίου της ΕΚΤ, δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή ε, επιτόκιο αναφοράς πέραν της ε, οριμότητας της επαύρων με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθούμε και με βάση έναν επαρκή αριθμό συναλλαγών. Άρα μπορεί να χρειαστεί για την παραγωγή αυτών των επιτοκίων να προβούμε σε μια κρίση, αλλά όχι εμείς, όχι μια κεντρική τράπεζα δηλαδή. Άρα πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος boring ε, με βάση τις ε, ισχύουσες συνθήκες των αγορών και μπορεί να προκύψει σύγκρουση ή ιδέα πως μπορεί να υπάρχει σύγκριση. Εάν μια κεντρική τράπεζα παρέμβει και θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής. Όχι, πρέπει να υπάρχουν λύσεις που θα δίνουν απάντηση ε, στις προκλήσεις εκείνες που μόνο ο τραπεζικός τομέας, ο ιδιωτικός τραπεζικός τομέας μπορεί να εντοπίσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, πρόεδρε. Χαίρομαι που σας έχουμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, πριν ολοκληρωθεί η θητεία. Θέλω να επανέλθω στη συζήτηση που έχουμε ξανακάνει αρκετές φορές. Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται την ιστορία του ευρώ. Λέτε ότι πρόκειται για κυριαρχία, ενίσχυση κυριαρχίας. Και θέλω να συμφωνήσω εδώ μαζί σας, γιατί πριν από το ευρώ είχαμε τους δύο μοχλούς, την δημοσιονομική και την οικονομική πολιτική, που κάλυπταν την ίδια γεωγραφική έκταση των χωρών μελών. Αποφασίσαμε λοιπόν λοιπόν να προχωρήσουμε την νομισματική πολιτική χωρίς όμως χρόνος να σπρώξουμε και προς την άλλη κατεύθυνση. Αν δηλαδή έχετε μια νομισματική πολιτική με ομοιογενή τρόπο, που συνήθως γίνεται, η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να είναι ικανοποιητική για ολόκληρη την επικράτεια, για ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό και χρειάζονται κάποια μέσα τα οποία θα επαναφέρουν την ισορροπία στην επικράτεια. Αν τώρα την νομισματική πολιτική την προχωρήσετε χωρίς να προχωρήσετε σε ένα βαθμό τη δημοσιονομική πολιτική, αυτό που κάνετε είναι ότι χάνετε κυριαρχία στη διαδρομή. Εγώ δεν βλέπω την διαδικασία ολοκλήρωσης σαν απώλεια κυριαρχίας, αλλά δεν βλέπετε σε επίπεδο Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, την ίδια ποιότητα κυριαρχίας που έχετε σε εθνικό επίπεδο. Δύο παράγοντες υπάρχουν τώρα εδώ πέρα. Ή που πάλι θα ξαναβρείτε τη συνοχή σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή θα βγείτε από το ευρώ, κάτι το οποίο δεν είναι δικιά μας πολιτική βέβαια, όπως είναι γνωστό, ή που θα προσθέσετε το κομματάκι που λείπει στον ομοσπονδιακό χαρακτήρα, δηλαδή έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης, συγχρόνως με την ικανότητα όμως ε, φορείς πράξης, προκειμένου να μπορεί κανείς να συλλέξει φόρους και να τους δαπανίσει. Εγώ εντάξει, σέβομαι τις απόψεις αυτών που λένε ότι το αντίθετο πρέπει να γίνει πριν να βγούμε από το ευρώ. Αλλά θέλω να ακούσω τις δικές σας σκέψεις επ' αυτού. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το οικοδόμημα που βασίζεται σε κανόνες μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του έτσι. Απάντηση. Δεν είναι εύκολη η ερώτησή σας. Πρώτον, ας κοιτάξουμε πρώτα την νομισματική πολιτική. Μέχρι τη συνθήκη του Μάστριχτ, κάθε χώρα ισχυριζόταν ότι είχε τη δικιά της νομισματική πολιτική. Μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες χώρες δεν είχαν καθόλου κυριαρχία επί της νομισματικής τους πολιτικής. Σωστά, η Γερμανία είχε. Και οι υπόλοιπε χώρες είχαν επιλέξουν είτε να κολλήσουν τα δικά τους τα επιτόκια σε αυτά των γερμανικών ή να υποτιμήσουν το νόμισμά τους. Κάποιες χώρες λέγανε ότι έχουν κυριαρχία πάνω στη νομισματική τους πολιτική, αλλά ακόμα και αυτές οι οποίες κάναν υποτίμηση τακτικά στο νόμισμά τους δεν είχαν ουσιαστικά κυριαρχία. Γιατί αν δεις πώς υπολογίζουμε αυτή την κυριαρχία που είναι η σταθερότητα των τιμών, ο πληθωρισμός, η απασχόληση, Αυτέ οι χώρες βρέθηκαν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από εκείνε οι οποίες συνέδεσαν ε, το δικό τους νόμισμα με εκείνο της Γερμανίας. Αυτή η κατάσταση Λοιπόν, ξεπεράστηκε όταν δημιουργήθηκε ο θεσμό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ακόμα και χώρε που δεν είχαν κυριαρχία πριν, είχαν μια πολύ χαλαρή κυριαρχία, δεν είχαν αξιοπιστία, ανάκτησαν κυριαρχία και αξιοπιστία. Στο δημοσιονομικό τομέα αυτή η ίδια πρόοδος θεωρήθηκε κάτι πιο δύσκολο, ας το πούμε έτσι, εξαιτία ε, της ίδιας της ουσίας των αποφάσεων των νομισματικών και του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις αποφάσεις αυτές του προπολογισμού, ε, που η άσκηση γινόταν στα εθνικά κοινοβούλια. Μπορεί κανείς να πει δηλαδή ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν γινόταν τόσο στη νομισματική πολιτική. Αλλά ιστορικά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή σε κάποιες ιστορικές περιόδους ναι, σε κάποιες όχι. Αυτή πάντως ήταν η κατάσταση. Αλλά ακόμα και έτσι οι κανόνες αποφασίστηκαν και επιλέχτηκαν. Βάσει του συστήματος κανόνων λοιπόν, πότε δεν χάνεις την κυριαρχία σου. Όταν οι κανόνες δεν είναι δεσμευτικοί. Όταν δεν είναι δεσμευτικοί ε, συνολικά κατά μέσο γιατί μερικές φορές φυσικά υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες, άλλες φορές όχι. Τότε μπορούμε να πούμε ότι η χώρα διατηρεί την κυριαρχία της. Πώς? Μια χώρα χάνει κυριαρχία όταν το χρέος της είναι ιδιαίτερα υψηλό. Όταν το χρέος είναι ιδιαίτερα υψηλό, δεν χρειάζονται καν κανόνες για να περιορίσουν την κυριαρχία της χώρας. Οι αγορές το κάνουν αυτό. Οι αγορές λένε στη χώρα τι αντέχει και τι δεν αντέχει η χώρα, τι είναι αξιόπιστο και τι δεν είναι. Οπότε η χώρα χάνει την κυριαρχία της η χώρα ή ο θεσμό οτιδήποτε, όταν το χρέος καταστεί τόσο υψηλό που οποιαδήποτε πολιτική δράση πρέπει να ελεγχθεί τελικά από τις αγορές. Δηλαδή από ανθρώπου που δεν ψηφίζουν, που βρίσκονται εκτός της ε, διαδικασίας δημοκρατικής λογοθεσίας. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η παρέτηση από την κυριαρχία. Αυτή είναι η ζωή. Και αυτό γίνεται από πολιτικές αποφάσεις που πήραν κατά το παρελθόν αυτές οι χρωμένε χώρες. Αυτό είναι ο λόγος. Τώρα, ποια είναι το φέλη των κανόνων. Είναι ότι αν υπάρξει συμμόρφωση, τότε προχωράμε στη σύγκληση. Και αυτό είναι το άλλο σκέλος της κυριαρχίας. Δηλαδή, σε ένα νομισματικό χώρο δεν είναι δυνατόν να έχουμε κυριαρχία εάν η οικονομία αποκλίνει συστηματικά αν η χώρα βρίσκεται πίσω σε ανταγωνιστικότητα, σε μεταρρυθμίσεις και επιπλέον έχει ιδιαίτερα υψηλό χρέο. Έτσι κινδυνεύει η κυριαρχία. Οι αιτίε για να χάσει κανεί κυριαρχία, σίγουρα συμφωνώ μαζί σα, έχουν να κάνουν με το πλαίσιο, με του κανόνε, το ότι περνάμε από του κανόνε, του θεσμού. Και αυτό εν μέρη αντιμετωπίζεται. Αλλά πολύ πριν το θέμα έχει να κάνει με τις πολιτικές. Η κυριαρχία απολύεται εξαιτία εσφαλμένων πολιτικών. Δεν χρειαζόμαστε έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης. Μια ερώτηση. Απάντηση. Μα πρόκειται για συνδυασμό. Το είπα και στην εισαγωγή μου. Διακόπτει ο πρόεδρος. Τι, μιλάω πολύ. Υπάρχουν και άλλοι. Πολύ σύντομα απαντήστε παρακαλώ σε αυτό γιατί είναι ενδιαφέρον και εντάξει θα κερδίσουμε το χρόνο στη συνέχεια. Εκτός μικροφώνου σχόλιο, δεν ακούγεται. Δεν ακούστηκε. Θα επανέλθουμε. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις προς την ίδια κατεύθυνση και θα μπορέσει ο κύριος Δράγκη να απαντήσει. Γκουέ δεν βλέπω, μόνο. Πρόεδρε. Πρόεδρε Δράγκη, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω ότι πολύ εκτίμησα τον νομισματικό διάλογο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, αλλά δεν είμαι και τόσο ενθουσιώδης για τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για το φέλη από το ενιαίο νόμισμα τα 20 τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματα κοινωνικά και οικονομικά στη χώρα μου, τη Γαλλία για παράδειγμα, είναι κακά και νομίζω και στη δικιά σας χώρα, την Ιταλία επίσης. Για κάτι άλλο θέλω να μιλήσω. 14 Δεκεμβρίου υπήρχε η διάσκεψη της Ευρωζώνης που ενέκρινε προτάσεις όσον αφορά το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και μεταξύ άλλων αναφέρεται η μεταρρύθμιση των ΚΑΚ που συμπεριλαμβάνονται στους ε, τίτλους του ευρώ. Πρόκειται για το Σύνταγμα που έχει να κάνει με την ε, μειοψηφία που αποκλεί μια απόφαση κλπ. Πρόκειται για μια προσπάθεια να γίνεται την διάρθρωση του χρέου πιο εύκολη. Μα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να έχει παραπάνω χρέο από μια χώρα από το όριο μπλοκαρίσματο για να μην πρέπει να ψηφίσει υπέρ μια αναδιάρθρωση. Το οποίο θα σήμαινε με τη σειρά του απευθεία αναχρηματοδότηση. Όμω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα έχουν 25% των χρεών τη Ευρωζώνη μετά από το τελευταίο σχέδιο. Προκειμένου να σταματήσει η ποσοτική χαλάρωση και να υπάρξει σταθεροποίηση του 25%, τι θα γίνει με τη μεταρρύθμιση των ΚΑΚ. Και το τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης έχει να κάνει με την προοπτική πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ή και με τη μεταρρύθμιση ακριβώς των ΚΑΚ. Δεύτερη ερώτηση όσον αφορά τα συμπεράσματα της διάσκεψης της Ευρωζώνης που προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα μπορεί να διαπραγματεύεται την αναδιάρθρωση με του ιδιωτικού πιστωτέ. Δεν πιστεύετε ότι αυτή η νέα διάταξη για κυρίαρχο χρέο θα δημιουργούσε πανικό στου επενδυτέ προκυκλικά και έτσι θα διευκόλυνε μία πάυση πληρωμών. Τα προνόμια του ταμείου αυτού δεν κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε αναταράξεις για την συνέχεια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Η απάντηση όχι. Γιατί αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε τις ε, αγορές στοιχείων ενεργητικού τον Ιούνιο, όχι επειδή προσκουράμε στα όρια που τους άλλους εμείς είχαμε ορίσει, Γιατί έχουμε περιθώριο. Το κύριο όμως στοιχείο αυτής της απόφασης ήταν ότι το απόθεμα που επιτύχαμε, το είπατε και στις 25% του συνολικού κρατικού μακροχρόνιου κρατικού χρέους της Ευρωζώνης είναι τόσο μεγάλο που οι καθαρές προσθήκες στο απόθεμα αυτό είχαν όλο και πιο μικρές, μικρό αντίκτυπο, αμεληταίο αντίκτυπο. Άρα ξέρουμε ότι με το απόθεμα αυτό που έχουμε μπορούμε πάντα να εξασφαλίζουμε το κίνητρο, το νομισματικό, που είναι απαραίτητο για την σύγκληση του προπληθωρισμού προς τους στόχους μας. Και αυτό που είδαμε επίσης τον Ιούνιο ήταν ότι τα επιτόκια, το έχω ξαναπεί, ε, κατέβηκαν, μειώθηκαν και έγιναν πιο ευνοϊκά συνολικά με τη δομή τους. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μας λένε ότι δεν οδήγησε σε νομισματικό περιορισμό, νομισματική περιστολή αυτή η απόφαση. Η δεύτερη ερώτηση. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Κοιτάξτε, ρητή εντολή για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο να αναλαμβάνει την αναδιαπραγμάτευση κρατικού χρέους δεν υπάρχει. Με πολύ προσοχή έχει διατυπωθεί ε, η φράση που λέω ότι θα πρέπει προς την κατεύθυνση αυτή να διευκολύνει κτλ. Ακριβώς για τους λόγους που εσείς αναφέρατε. Βεβαίως και είναι πρόβλημα το να υπάρχουν υψηλά ποσοστά χρέους σε ορισμένε χώρε, αποθέματα χρέους. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη και τη νομισματική σταθερότητα, γιατί δεν θέλουμε το φάρμακο να είναι χειρότερο. Και βεβαίω τα αποθέματα αυτά χρέους μπορεί να είναι και 20 αιτίε και πιο παλιά ακόμη. Άρα, με ένα πολύ προσεκτικό, επιφυλακτικό τρόπο έγινε η απόπειρα ουσιαστικά να πούμε πώς το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο μπορεί να αναλάβει ρόλο εκεί όπου μπορεί γενικά να γίνει μια συζήτηση για να διαπραγμάτευση, αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτηκε κανείς πως θα μπορούσε το ΕΝΤ να προξενήσει αναδιαπραγμάτευση χρέους. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο μπορεί να διευκολύνει ε, συνομιλίες για χρέος κρατικό. Εάν μια χώρα που είναι σε πρόγραμμα αποφασίσει να προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση του χρέους της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κύριε Χιούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ και λέω ότι είναι πολύτιμη πηγή γνώσεων κάθε φορά που συναντιόμαστε τα λόγια σας. Και συνεχίζω με το ζήτημα αυτό των αγορών στοιχείων ενεργητικού και την μετακύληση στις επανεπενδύσεις. Μιλήσατε και για την ε, λογική που σα οδήγησε στην επιλογή αυτή. Ρωτώ όμω, εάν σωστά αντιλαμβάνομαι πως ε, τώρα στην τρέχουσα περίοδο λαμβάνετε υπόψη διαφορετικέ παραμέτρους για τις αποφάσεις που λαμβάνετε. Άλλες από αυτές ε, που ακολουθούσατε στο πρόγραμμα αγοράς ή στα χρόνια που λειτουργούσε το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού έχει αλλάξει κάτι άλλο ή έστω η στα χρόνια που λειτουργούσε το πρόγραμμα αγορά στοιχείων ενεργητικού. Έχει αλλάξει κάτι άλλο ή έστω η ένταση των ε, ε, στοιχείων που λαμβάνει την υπόψη. Και δεύτερον, μπορείτε ανατρέχοντας την περίοδο αυτή της προσωπική χαλάρωσης να επισημανετε κάτι το επικριτικό ή ότι ο μηχανισμός για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής έχει εντωμεταξύ τροποποιηθεί, έχει εξελιχθεί από την περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης. Ευχαριστώ. Δράγκη. η διακοπή του προγράμματος ε, αγοράς ενεργητικού που όπως είπα ήταν ε, ότι σταθεροποίησε τελικά το απόθεμα χρέους δεν οδήγησε όμως σε μείωση χρέους είπαμε ότι υπήρξε μια εναλλαγή των εργαλείων από την αγορά στοιχείων ενεργητικού. Έχουμε περάσει τώρα στην ε, καθοδήγηση, forward guidance, ε, επιτόκια δηλαδή και συζήτηση με όποιον ε, μας ρωτάει, όπως μας ρώτησαν ε, κατά το τέλος του προγράμματος ε, στοιχείων ενεργητικού, πότε θα μειώσετε το μέγεθος του ε, ισολογισμού όπως το πράττει ήδη η ΦΕΔ επί παράδειγμα, Εμείς λοιπόν είπαμε ότι περιορίζουμε τον ορίζοντα σε σχέση με την πιθανότητα αύξησης ή μετακυλίουμε τον ορίζοντα σε σχέση με την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων για μετά το καλοκαίρι και από εκεί μπορούμε να δούμε αν υπάρχει λόγος να ε, συνεχίσουμε. Άρα έχουμε μια κυλιόμενη χρήση των ε, εργαλείων. Τώρα, απόδειξη της διευκόλυνσης στην ε, επίλυση της κρίσης που προσέφερε η ποσοτική Χαραλός, νομίζω ότι είναι συντριπτική και προφανής. Αν πάρουμε σαν ε, σημείο αναφορά χρονική το 2014 και κοιτάξουμε την περίοδο τότε, έχουμε μακρό, μακρό κατάλογο δικτών και χρονικά που μας δείχνει σε ποιο βαθμό η ποσοτική χαλάρωση βοήθησε και για τα επιτόκια και για το δανεισμό των τραπεζών μέχρι και στοιχεία που μας λένε ότι στην περίοδο 2016-2019 η ποσοτική χαλάρωση και μόνο είχε συμβολή στο 1,9% ε, στον πληθωρισμό σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αλλά αυτές είναι στατιστικές τι οποίες δεν θα ήθελα να δώσω πολύ μεγάλο βάρος. Απλώς νομίζω αποτελούν ένα στιγμιότυπο της Κατάσταση Πάντως κάθε πτυχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος μόνο με την, ε, τον κατακαιρματισμό που γνωρίζαμε το 2014 που μειώναμε διαρκώ τα επιτόκια χωρίς ανταπόκριση από τις τράπεζες σε χαμηλότερα επιτόκια σε ορισμένε. Ε, δανεισμού. Σε ορισμένε χώρες μπορεί, ναι, να μειώνονταν, αλλά ήταν πολύ κατακαιρματισμένο ο χρηματοπιστωτικό κόσμο. Ε, ε του ίδιου ομίλου ε, σε χώρες διαφορετικές, μία του κέντρου, του πυρήνα, του σκληρού πυρήνα του ευρώ και άλλη της, του, περιφέρειας, ε, έπαιρναν διαφορετικές αποφάσεις σχέση με τα επιτόκια δανεισμού. Αυτό λοιπόν χάρη στην ποσοτική χαλάρωση αλλά και σε άλλες νομισματικές πολιτικές που έχουμε αναλάβει, όχι μόνο την ποσοτική χαλάρωση, είδαμε ότι έχουν μετατραπεί πια σε μια πολύ μακρινή ανάμνηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνκ. Ευχαριστώ και εσά κύριε Πρόεδρε και εσά κύριε Πρόεδρε Ντάγκη. Ε, ευχαριστώ για την παρουσία σα εδώ. Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης πάντοτε είναι θέμα που συζητείται. Λέτε επίσης και πολλοί κεντρικοί τράπεζες ότι η Ευρωζώνη από την μια μεριά το ε, ο κίνδυνος ε, ιδιωτικών ε, πτωχεύσεων ιδιωτών στις ε, ΗΠΑ είναι πολύ περιορισμένος. Εδώ πέρα φαίνεται πως αυτό παίζει ένα σημαντικότερο ρόλο. Η Κεφαλαιακή Ένωση έχει συμβάλει στην ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Τώρα, για την χρηματοδότηση. Άκουσα τον Μπερνά Κερέ να λέει ποιο είναι ο ρόλο για την ανθεκτική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Και αν θέλουμε να αλλάξει κάτι εκεί, οι επόπτες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και ιδίως βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι και ζήτημα ανθεκτικότητας. Γιατί χρειαζόμαστε μια μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια μέσα από ε, σοκ, από διαρκή σοκ. Πώς βλέπετε, θεωρείτε δηλαδή ότι η κίνδυνη που συνεπάγεται μια πολιτική για την αντιμετώπιση του αλλαγής του κλίματος ενδέχεται να μας οδηγήσει σε ε, δυσχερή και ανηφορικό δρόμο προς την ε, κατεύθυνση της ε, Κεφαλαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος Δάκη, σας ευχαριστώ. συμφωνώ μαζί σας στο εξή. Η Κεφαλιακή Ένωση και η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα έχουν δύναμη από την άποψη της, ε, του, της μοιράσματος των, των κινδύνων γιατί θα καταστήσουν μικρότερο τον κίνδυνο για τον προπορισμό. Αν μπορεί δηλαδή να είναι δυνατόν να απορροφήσουν τους κραδασμούς, ε, βλέπετε ότι από τις πραγματικές ε, χρηματοπιστές αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες απορροφώνται πολύ λιγότεροι κράδασμοι και αντιθέτω, πολύ μεγαλύτερο μέρος στην, ε, στην Ευρωζώνη απορροφάται από τους εθνικούς κράδασμους, πολύ περισσότερο από ό,τι στις ΗΠΑ ή σε άλλες ε, περιοχές με ένα νόμισμα. Άρα, η σε αλλες ε περιοχες με ενα νομισμα αρα η προοδο θα είναι αργή. Κάτι που φαίνεται ωστόσο να γίνεται όλο πιο σαφές και όλο και λιγότερο αποδεκτό είναι να μην γίνεται καμιά δράση σε κανένα από τα μέτωπα. Εγώ θέλω να δω να προχωρεί η Τραπεζική Ένωση και η Κεφαλαϊκή Ένωση. Εύκολο είναι βέβαια να πει κανεί ότι υπάρχουν πολιτικά θέματα και πολιτικά προβλήματα. Και βεβαίω εμεί οι κεντρικοί τραπεζίτε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λέμε. Διότι Αυτά είναι πολιτικές, ε, σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Υπάρχει όμως μια καθαρή γραμμή που επιβάλλει δράση. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση κινδύνων και σε καταμερισμό των κινδύνων. Και εκεί σωστό είναι να βρεθεί ο σωστός ρυθμός. Η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου έδειξε κάποια πρόθεση για μια κατεύθυνση προς τα εκεί. Έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα έχουν δοθεί κάποιες εντολές για να διεξαχθούν άλλες μελέτες για ορισμένα θέματα. Υπάρχει λοιπόν μια κίνηση. Εμείς θα ευχόμασταν να είναι ταχύτερη κίνηση αυτή, αλλά θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Αλλά ωστόσο να διατηρούμε τις ελπίδες μας. Τώρα για την αλλαγή κλίματος. Είναι σαφές ότι καθώς προχωρούμε κίνδυνοι που απορρέουν από την αλλαγή του κλίματος γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Όλο και πιο εμφανείς, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν έστω και μια πενταετία πριν. Ας δούμε όχι τόσο τον τραπεζικό τομέα, αλλά τον τομέα των ασφαλίσεων. Οι ασφαλίσει, οι ασφαλιστέ αντιλαμβάνονται πολύ εντονότερα του κινδύνου από την αλλαγή του κλίματο από ό,τι πριν από μια πενταετία. Άρα θα γίνει κάτι, θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάζουν οι επόπτε. Να πει κανείς ότι θα είναι εύκολη μετάβαση. Νομίζω ότι χρειάζεται και μια πολιτισμική αλλαγή που πρέπει να επέλθει. Άρα όλοι πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κερέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βέρνερ Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. επιθυμώ να επαναλάβω τους επένους και να τους συμπληρώσω που ακούσατε από άλλους συναδέλφους. Περάσατε και δύσκολες στιγμές εδώ στον ε, νομισματικό διάλογο, σας επέκριναν και πολύ. Μπορεί να πει κανείς σήμερα ότι το ευρώ είναι επιτυχία. Όταν ο Greenspan εμφανίστηκε στο Κογκρέσο, στην Βουλή των Αντιπροσώπων και είχε δηλώσει ότι θα αποτύχει το ευρώ. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η πρόβλεψή του αποδείχθηκε εσφαλμένη. Τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Είπατε πριν ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εθνικές μεταρρυθμίσεις, τα project και να μειώσουμε τους κινδύνους. Έχω τώρα τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής. Εφόσον αμφισβητείτε ξανά και ξανά, τι έχετε να προτείνετε, πρόσθετες αρμοδιότητες θα πρέπει να αναλάβει ο Επίτροπος Αρμόδιος για τα Δημοσιονομικά. Δεν θα αποκτήσουμε Ευρωπαίο Υπουργό ε, Δημοσιονομικών ή Οικονομικών καλύτερα. Οπότε αυτός ο Επίτροπος τι θα πρέπει να αναλάβει στο χαρτοφυλάκιο, του. Δεύτερη ερώτηση η κατασκευή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης μπαίνει στο πακέτο των μεταρρυθμίσεων. Έχει αμφισβητηθεί κατ' επανάληψη το ότι ε, κάθε χώρα μέλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν πάει ανάλογα με την οικονομική δύναμη των μελών. Μπορείτε να πείτε κάτι σχετικά. Τρίτο, λόγω των διαθροτικών προβλημάτων και των διεθνών αναταράξεων, πολλοί επιστήμονες έχουν πει ξανά και ξανά ότι ο δρόμος προς τα πίσω από τα προγράμματα αγοράς ε, στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή κατεύθυνση Fed ή προς τα μπρος κατεύθυνση Ιαπωνικής Κεντρικής Τράπεζας που δεν αντιμετωπίσει κανένα περιορισμό σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να αγοράζει μετοχές, ε, ε, μετοχές επιχειρήσεων που ενδεχομένω να αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Δεν είμαι βέβαιο ότι κατάλαβα καλά την πρώτη σα ερώτηση να, να κάνω μια σύντομη συμπλήρωση. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν ο Επίτροπος Αρμόδιος για τα νομισματικά θα πρέπει να αναλάβει στο χαρτοφυλάκιό ό,τι περισσότερες αρμοδιότητες, διότι οι χώρες μέλη δεν τηρούν αυτά τα οποία έχουν οι ίδιες υπογράψεις ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές τους δεσμεύσεις. Σας ευχαριστώ. μου θέτετε μια ερώτηση. Εγώ με κάπως ε, κλείνω προς μια ε, απάντηση, αλλά θα απαντήσω πρώτα στη δεύτερη σα ερώτηση. Με ρωτάτε αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αποτελέσει, να μπει μέσα, σε αυτή, μέσα και αυτή στο πακέτο μεταρρυθμίσεων για το μέλλον. Όπως είπα, ε, επ' αυτού δεν είμαι αντικειμενικός παρατηρητής. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το παρόν καθεστώς. Και θεωρώ ότι αν πρόκειται να ξανανοίξουμε μια συζήτηση για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα το κάναμε αυτό, αλλά υπό δύο όρους. Ο πρώτος είναι ότι το Ευρωπαϊκό, Κεντρικό, το Ευρωπαϊκό μάλλον Δικαστήριο να έχει διαπιστώσει ότι έχουμε παραβιάσει το καθεστώ, το καταστατικό μα δηλαδή, ή να βρει λόγου για του οποίου θα έχουν αλλάξει, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχουμε δει. Και το άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην έχει ανταποκριθεί εντολέ τη υπό το παρόν καταστατικό τη. Αλλά ελπίζω ότι ούτε αυτό συμβαίνει. Άρα δεν μπορώ να αποκλείσω κάποια εξέλιξη στο μέλλον. Αλλά επί του παρόντος φαίνεται να είμαστε πολύ απομακρυσμένοι από οποιαδήποτε νέα συζήτηση περί τροποποίησης, αναθεώρησης των συνθήκων τουλάχιστον του μεγέθου που υπονοείται. Τώρα για την πρώτη σα ερώτηση, Ποιο είναι ο επίτροπο για τα νομισματικά, Currency Commissioner. Α, ναι, ναι, τώρα κατάλαβα. Άκουσα Currency Commissioner και δεν κατάλαβα καλά τι εννοείται. Κοιτάξτε, Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου αν εξετάσουμε τα τελευταία 20 χρόνια και συγκρίνουμε πώς απέδωσε η ε, ενσωμάτωση της νομισματικής πολιτικής και, με τις δημοσιονομικές πολιτικές. Θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι ότι η πρώτη απέδωσε καλύτερα από την δεύτερη, νομισματική από τη δημοσιονομική δηλαδή. Τώρα, προς τα εκεί προχωρήσαμε Πώς λειτουργούν τώρα οι θεσμοί, αυτό είναι ανοιχτό ερώτημα και μεγάλο ανοιχτό ερώτημα. Ορισμένοι εξημών, λοιπόν, είμαστε πεπισμένοι ότι βρισκόμαστε στο σημείο του τέρματος. Αλλά κανείς από μας δεν μπορεί να γνωρίζει απολύτως πώς θα λειτουργήσει η διακυβέρνηση των θεσμών αυτών. Αλλά να προσθέσω ένα πράγμα, το οποίο είναι σχετικό, διότι όταν εξετάζουμε πώς λειτουργεί το Eurogroup, πώς προχωρεί δηλαδή στις συζητήσεις προϋπολογισμών εκατέρωθεν, αλλά και τα σχέδια προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εξέταση των μέτρων εκ των προτέρων στην διάρκεια των συζητήσεων, αλλά και εκ των υστέρων. Δεν είμαστε και τόσο μακριά δεν είμαστε και τόσο μακριά από το να θεωρηθεί το Eurogroup ως ένα εμβριώδες τέτοιο θεσμικό όργανο. Αυτό ε, μόνο ε, μπορώ να πω για την ώρα, γιατί το θέμα βέβαια είναι ευρύτατο. Thank you. Ευχαριστούμε. Πέτερ Σάιμον. Πέτερ Σίμον. Ε, αξιότιμε και Ντράγκη, Έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα για τα τελευταία 20 χρόνια καθώς και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσεως. Θέλω να πω και εγώ το δικό μου. Να σας πω κάτι το οποίο έχω πει κάποτε σε προσωπική συζήτηση μαζί σας, ότι είναι πεποίθησή μου, ότι αν εσείς τότε που οι πολιτικοί στις πρωτεύουσε δεν ήταν σε θέση να ασκήσουν πολιτική, αν εσείς ως μοναδική προσωπικότητα δεν είχατε ασκήσει τότε πολιτική δεν θα είχαμε διασώσει το ευρώ. Και γι' αυτό σας είμαστε όλοι εδώ πραγματικά ευγνώμονες. Έχω να πω, έχω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την οποία ε, θέσατε ως εναλλακτική επιλογή, εάν δεν θέλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκός προπολογισμό. Δεν το είπατε ακριβώ έτσι, αλλά είπατε ότι πρέπει κανείς να αποφασίσει. Θέλει κοινό ευρωπαϊκό προπολογισμό ή θέλει τραπεζική ένωση βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η εμπιστοσύνη των χωρών μελών, των μεν προς τις δε, δυστυχώ μειώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αν δούμε τι χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση, εσείς μιλείτε για παράδειγμα για την ενία ε, ε, εγγύηση καταθέσεων, που δεν υπάρχει ακόμη. Αλλά αυτό που λείπει είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών. Εάν σκεφτούμε τώρα πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη αυτή. Υπάρχουν κατά την άποψή σας κάποιοι δρόμοι που δεν έχουμε ακόμη ακολουθήσει, αλλά που θα έπρεπε να συζητήσουμε. Κάποτε συζητούσαμε για ενδεχόμενη ε, μείωση του χρέους. Έπαυσε αυτή η συζήτηση. Τι άλλους εναλλακτικούς δρόμους μπορούμε να ακολουθήσουμε, ώστε πέρα από κυρώσεις να μπορέσουμε να κυρώσουμε την των, ε, δηλαδή, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε παροχή κινήτρων ώστε όλοι να συμβάλλουν. Συμφωνώ μαζί σας και νομίζω ότι το έχω πει και άλλες φορές. Εμπιστοσύνη και σύγκριση είναι οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η πρόοδος για την εμβάθυνση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η σύγκριση μπορεί να επιτευχθεί με οικονομική ανάπτυξη αλλά και με διαφθορτικές μεταρρυθμίσεις. Και τα δύο πράγματα. Α το πω διαφορετικά, ο καλέ και αν είναι οι προθέσει, δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη αν δεν υπάρχει σύγκληση. Εάν η χώρα μέλο γίνεται όλο και ασθενέστερη, και οι δύο πυλώνες δηλαδή πρέπει να υφίστανται. Εάν περιορίσουμε, αν στρέψουμε την προσοχή μας μόνο σε ε, πολιτικές δράσεις, η εμπιστοσύνη ανακτάται, αποκτάται ή ανακτάται αναλόγως, με την αντιμετώπιση των διαρκών θεμάτων που έχουν καταστήσει τόσο δύσκολη την ε, πρόοδο, όπως το NPL, όπως ε, ε, τα asset επίπεδο 3 και 4, το επίπεδο του χρέους σε ορισμένες άλλες χώρες, το δημόσιο χρέος στους ισολογισμούς άλλων χωρών. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά θα πρέπει και να συνοδευτούν, να συνοδεύονται από ξεκάθαρα ορισμένη πολιτική οδό που να ακολουθηθεί θα πρέπει να συνοδεύονται από καλές προθέσεις και από ανάληψη δεσμεύσεων για να προχωρήσουν οι χώρες σε ένα risk sharing, σε ένα καταμερισμό κινδύνων. Τα δύο πράγματα πηγαίνουν χέρι με χέρι και θα πρέπει να υπάρξει και ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα όπου θα συμβούν τα διάφορα βήματα και μάλιστα με συγκεκριμένα νούμερα. Υπό την έννοια αυτή, η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου έδωσε κάποια όθηση. Υπάρχει και μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου που έχει λάβει την εντολή να ε, ασχοληθεί με το ίδιο, e με τις ασφαλίσεις και έχει γίνει δεκτό το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί ευρεία εντολή και σε ό,τι αφορά την Κεντρική Τράπεζα, το απότατο τέλος θα πρέπει, τις διαδικασίες αυτής, θα πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο να είναι αμοιβαίο μεταξύ των χωρών μελών. Θα χρειαστεί πολλούς χρόνο για να φτάσουμε εκεί, αλλά και στον τομέα αυτό, όπως και σε πολλούς άλλους που αφορούν το βάθεμα της ε, νομισματικής Ένωση χρειάζεται ένα ξεκάθαρο τέρμα. Αυτό θα δώσει μεγάλη ενεργητικότητα και στις δύο πλευρές, και για την μείωση των κινδύνων, αλλά και για, την, για τον καταμερισμό των κινδύνων. Αυτό πρέπει ε, να είναι ο στόχος και των δύο πλευρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρτουσέλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Ντράγκη, θέλω να σας ευχαριστήσω ως Ιταλός, διότι μας κάνατε περήφανος που είμαστε Ιταλοί. Και μάλιστα μια χώρα που έχει ανάγκη από ηγετικά στελέχη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μας κάνατε να αισθανθούμε περήφανοι και που μας στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ρωτήσει λοιπόν. Πρώτον για την κατάσταση στη χώρα μου, η Banca d'Italia, η Ιταλική Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Ορματικό Ταμείο μετά, είπαν ότι φαίνεται να διαγράφεται μια σαφής επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. 1% προβλέπει η κυβέρνηση, 0,6% μας λένε. Και Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τονίζει τους κινδύνους από το χρέος περιγράφοντας μια κατάσταση που θα οδηγούσε και σε μείωση της ανάπτυξης. Ενώ σήμερα ο Υπουργός Σαββόνα ενώπιον της ε, Βουλής της Ιταλικής είπε ότι τα εργαλεία με τα οποία έγινε αυτός ο υπολογισμός είναι πεπαλαιωμένα και ότι πρέπει να γίνει πιστευτός εκείνος ο οποίος ως καθηγητής είναι πιο αρμόδιος για να ε, δώσει προβλέψει από το Διεθνές Σωματικό Ταμείο. Ωστόσο, θεωρώ ότι φαίνεται πως πρέπει να προετοιμαστεί για ένα διορθωτικό προπολογισμό η Ιταλία, καθώ βλέπουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ε, προεξαγγελθεί δεν υλοποιούνται και πρέπει να προχωρήσουν. Πρώτο αυτό. Σε σχέση με την ε, έκδοση του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ. Αποφασίστηκε η πάυση αυτής της, ε, αυτού του, τραπεζογραμματίου, πάυση έκδοσης του για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Ωστόσο, μήπως θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μια ε, παράλληλη δράση ελέγχου πέραν του να σταματάει δηλαδή, το, το, το τραπεζογραμμάτιο, να υπάρχει και ο έλεγχος στα τραπεζικά ιδρύματα. Ο κύριος Δράκη, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την Ιταλία. Η κατάληξη του διαλόγου με την Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό ήταν νομίζω θετική είδηση. Είπατε ότι το ε, spread μειώθηκε ελαφρώς. Άρα ο διάλογος και η συμμόρφωση στους κανόνες οπωσδήποτε έχει θετικό αντίκτυπο στο spread και τις δυνατότητες για χρηματοδότηση για τους πάντες. Το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είπα και νωρίτερα, δεν θα είναι τόσο ε, ζωτικό, δεν θα είναι τόσο ζωντανό όσο πριν και βλέπουμε ότι η Ιταλία δεν έχει την ανάπτυξη που είχε στο παρελθόν. Αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι αρχικά έχει υπολογιστεί η ανάπτυξή της και αυτό νομίζω το βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιο έντονα στην Ιταλία. Πάντα όμως όταν, ε, και στην ανάπτυξη, όταν είχε ανάπτυξη ευρωζώνη, η Ιταλία πάλι είχε χαμηλότερη ανάπτυξη από άλλες χώρες. Άρα ίσως είναι πρόημο να μιλήσουμε για διορθωτικό προϋπολογισμό. Ίσως θα πρέπει να δούμε και τα επιμέρους στοιχεία του προϋπολογισμού. Ε, στοιχεία δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή ακριβή για το πώς θα υλοποιηθεί και τι συνέπειες θα έχει. Πρέπει να δούμε και τα φορολογικά έσοδα, εάν θα έρθουν όπως θα προβλέπουν. Για τα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ. Θα θυμάστε ίσως ότι στις 4 Μαΐου του 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε πως το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα αποκλειστεί από τη σειρά Europa και θα σταματήσει η έκδοσή του προς τα τέλη του 18, αρχές του 19. Τώρα, οι εθνικές τράπεζες θα μπορούν να διαθέτουν τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ στους πελάτες τους μέχρι τις 26 Ιανουαρίου του 19. Τώρα γιατί να είναι φυσιολογικό αυτό. Ε, ας σκεφτούμε ποιοι είναι οι χρήστες των τραπεζογραμματιών των 500 ευρώ. Υπάρχουν περιοχές του κόσμου που με μεγάλη χαρά εισπράττουν το 500 Γιατί ενώ κάπου θεωρείται ε, ευλογία η διακοπή της εκδοσής του, ενώ αλλού ε, προξενεί ανησυχίες, νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε. Στη μετάβαση τώρα, η Bundesbank και η Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας εκδίδουν τραπεζογραμμάτια μέχρι τις 26 Απριλίου του 2019. Αφού σταματήσει η έκδοση, το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ, ευρώ παραμένει νόμιμο, νομισματικό ε, συνάλλαγμα. Επομένως θα έχει την ονομαστική του αξία, δεν τη χάνει. Αυτή είναι η απάντησή μου το αντιμετωπίζουμε όπως κάθε άλλο ε, τραπεζογραμμάτιο. Όχι εμείς, δηλαδή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, θα σας υποβάλω δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Η μία αφορά τα κόκκινα δάνεια τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε στην Ελλάδα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατασχέσεις και πληστηριασμών κατά των Ελλήνων οι οποίοι έχουν φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια. Ούτε βέβαια αποτελεί λύση το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες σε διάφορα funds, τα επωνομαζόμενα κοράκια, σε εξευτελιστικές τιμές. Επανειλημμένα έχω προτείνει να δημιουργηθεί ένα ταμείο σωτηρίας δανειοληπτών ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ μέρους του ελληνικού κράτους προκειμένου να αγοράσει τα κόκκινα δάνεια στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα funds, δηλαδή περίπου κάτω από το 10% της αξίας τους. Και εν συνεχεία να καλέσει τους φτωχοποιημένους δανειολήπτες να εξοφλήσουν τα δάνειά τους στο ίδιο ποσό. Πώς θα έβλεπε αυτό το σχήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς από τη μια θα υπήρχε η προστασία των δανειοληπτών που πράγματι αδυνατούν να πληρώσουν και αφετέρου θα υπήρχε απαλλαγή των τραπεζών από κόκκινα δάνεια ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την ε, ποσοτική χαλάρωση. Η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από την ποσοτική χαλάρωση, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, συμμετέχει στην ποσοτική χαλάρωση και έχει πληρώσει μέχρι το 2017 62 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημά μου είναι πότε θα εντάξετε τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στην ποσοτική χαλάρωση. Είχατε πει τον Ιούνιο ότι ο ίδιος ως Κεντρική Τράπεζα θα κάνατε τη δικιά σας έρευνα και έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Έχετε ολοκληρώσει αυτό. Και δεύτερον, πότε θα δοθεί η δυνατότητα ομόλογα των ελληνικών εταιριών να ενταχθούν και αυτά στην ποσοτική χαλάρωση και να μπορούν να αγοραστούν από τις κεντρικές τράπεζες ή και από την ε, Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή την Ελληνική Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ. Thank you. The... Ευχαριστούμε. Να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση. Θα το κάνουμε όταν γίνουν επιλέξιμα. Τώρα δεν είναι. Έχουμε κριτήρια και βρίσκονται κάτω από αυτά τα κριτήρια. Για το πρώτο, Γνωρίζουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σχολιάσω πραγματικά, γιατί όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Όμως, μειώνοντας ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάποιοι από αυτούς που έχουν τα χρέη αυτά αποτελούν ε, μέρος ενός μεγαλύτερου, πολύ ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος και από την άλλη μεριά έχουμε και τους στρατηγικούς δανειστές. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Αλλά αντιμετωπίζοντας τους πιο φτωχούς δανειολήπτες, Υπάρχουν δύο τρόποι για να αναβληθεί το πρόβλημα και να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα για τις τράπεζες. Οπότε οι τράπεζες στη συνέχεια δεν θα είναι σε θέση να δανείσουν ή να στηρίξουν το πρωτογενή τομέα όπως θα έκαναν αλλιώ. Το άλλο είναι να απαλλαγούμε. Δηλαδή να διατηρήσουμε τις πληρωμές, οπότε δεν θα επηρεαστούν οι τράπεζες αλλά θα βοηθήσουν απευθεία τους πιο φτωχούς δανειολήπτες. Νομίζω ότι έχει υπάρξει σημαντική... Νομίζω ότι έχει υπάρξει τέτοια προσπάθεια και οι ελληνικές τράπεζες μην ξεχνάμε ότι μόλις βγαίνουν από μια μακρά περίοδο που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν και να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα υπάρχει κεφαλοποίηση, τώρα μπορούν να στηρίξουν πραγματικά την οικονομία και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην τις επηρεάσουμε αρνητικά για το μέλλον. Έχω δέκα δευτερόλεπτα, ρωτάει ο κύριος Μαριάς. Απάντηση έχετε το χρόνο αργότερα. Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Τράγκη, υπάρχει μια καθοδική πορεία στην οικονομία από ό,τι λένε οι προβλέψεις σας παραμένετε με εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει μεσοπρόθεσμα να συγκλίνει. Όμως παρόλα αυτά υπάρχει μια επιβράδυνση και η οικονομική ανάπτυξη είναι πιο αδύναμη από το αναμενόμενο. Οπότε η προφανής ερώτηση είναι τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε γι' αυτό. Και όχι μόνο βέβαια να προσευχόμαστε. Οπότε άκουσα την απάντησή σας για την νομισματική πολιτική. Είπατε ότι η νομισματική πολιτική παραμένει υποστηρικτική επαρκώς και αν χρειαστεί θα γίνουν και περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως, κατά τα άλλα, έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τους πολιτικούς κινδύνους, ξεκινώντας από το Brexit. Θα συμφωνούσατε με την Βρετανική Κεντρική Τράπεζα ότι το σενάριο της έλλειψης συμφωνίας είναι το χειρότερο. Μας μένουν 8 εβδομάδες μέχρι το Brexit κανονικά. Οπότε εσείς θα λέγατε ότι το, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης είναι να φροντίσουμε να αποφύγουμε αυτό το σενάριο όπου δεν θα υπάρχει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερον, για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επισκόπησή της για το 2018 ζητάει περισσότερες επενδύσεις ποιότητας και πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική στις χώρες που έχουν αποθεματικό. Εσείς θα συμφωνούσατε για την ποιότητα των επενδύσεων και για την επεκτατική πολιτική στις πλειονοσβατικές χώρες, ότι αυτά θα φτάνανε για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να σταματήσει η επιβράδυνση. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας όσον αφορά το Brexit. Δεν είμαι και πολύ πρόθυμος να απαντήσω γιατί δεν θέλουμε ποτέ να παρεμβαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία είναι ήδη αρκετά περίπλοκη από μόνη της. Και επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Εμείς παρακολουθούμε, συνεργαζόμαστε με την Κεντρική Τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου, προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τις ε, αγορές έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο και έχουμε κάνει πολλή δουλειά μαζί τους. Έχουμε ομάδα εργασίας που λειτουργεί εδώ και αρκετούς μήνες. Οπότε πέρα από αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τα υπέρ και τα κατά των διαφορετικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της συζήτησης που λαμβάνει η χώρα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, η δικιά μας αρμοδιότητα είναι κατά κύριο λόγο να διασφαλίσουμε ότι όσον μας αφορά, εμείς έχουμε εντοπίσει τις δυσκολίες στην περίπτωση του κάθε σεναρίου και ότι έχουμε εντοπίσει τι δράση θα χρειαστεί στην κάθε περίπτωση. Πολλές από αυτές τις δυσκολίες και τα ενδεχόμενα μπορεί να μην χρειάζονται κάποια παρέμβαση και να φτάσει ο ιδιωτικό τομέα για να βλύνει τι συνέπειε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Υπάρχουν πολλά σενάρια, σύμφωνα με τα οποία είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι θα κάνουμε. Και σίγουρα η πρόσφατη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ισοδύναμα ήταν κάτι το οποίο βοήθησε πολύ. Τώρα έρχομαι στο, στη δεύτερη ερώτησή σας. Ναι, συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητούμε πολύ για το μέγεθος του προπολογισμού στις διάφορες χώρες. Μιλούμε πολύ λιγότερο, γιατί είναι πιο δύσκολο να το κάνουμε, για το ε, πόσο φιλικός προς την ανάπτυξη πρέπει να είναι κάθε φορά ο προπολογισμό. Το και 7-8 χρόνια πριν από την κρίση. Σε πολλές χώρες το έχουμε δει μια σημαντική αύξηση στις τρέχουσες δαπάνες και πολύ μεγάλη μείωση των δημοσίων επενδύσεων και μεγάλη αύξηση των φόρων. Οπότε δεν είναι περίεργο. Όταν μας έφτασε η κρίση, οι χώρες εκείνες που ακολουθούσαν αυτού του είδους την πολιτική η οποία ήταν ε, πολύ υπέρ της ανάπτυξης, ήταν πιο ευάλωτη στην κρίση. Επιπλέον, έχοντας συσσωρεύσει μεγάλο χρέος, το οποίο επηρεάζει τη δημοσιονομική πολιτική, περιορίζει και τα περιθώρια να αντιδράσει κανείς στην κρίση. Οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε στην σύνθεση του προπολογισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Τώρα το δεύτερο κομμάτι των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συμμετρική εφαρμογή της διαδικασίας ανισορροπιών. Και συμφωνούμε και σε αυτό. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Να δούμε τι σημαίνει. Τι σημαίνει για μια χώρα η οποία έχει πλήρη απασχόληση και εδώ μάλιστα και αρκετά χρόνια και ξαφνικά δεν έχει αρκετή απασχόληση, επεκτείνοντας μεγάλα τμήματα της οικονομίας της και να προτείνουμε ότι πρέπει να προβεί σε μεγαλύτερες δαπάνες. Είναι μια σωστή ερώτηση αυτή. Σίγουρα, αν αυτό σημαίνει επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, στην τεχνολογία, στις υποδομές, όπου χρειάζονται οι δαπάνες, αυτό είναι καλό, αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, γιατί πρέπει να αναρωτηθούμε οι περισσότερες αυτές δαπάνες πώς υλοποιούνται και πώς οι περισσότερες δαπάνες στις χώρες ε, τις πλεονασματικές θα έχουν επιπτώσεις δευτερογενώς και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Δεν είναι προφανής η απάντηση σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κλίντς ρωτήσα, σας ρώτησαν, σας έκανα άλλες, αρκετές δύσκολες ερωτήσεις, έχω δύο απλές. Πρώτη, την ιδιότητα μέλους της Ευρωζώνης. 26 από τις ακόμα 28 χώρες έχουν δηλώσει και υπογράψει ότι θα γίνουν κάποτε Ευρωζώνες. Από αυτές 7 δεν είναι ακόμα, αν και ορισμένες, μια ή δυο, ε, ανταποκρίνονται στα κριτήρια για να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη αυτή. Τη θεωρείτε ευκταία ή ίσως και αναγκαία αυτές οι χώρες μέλη, οι οποίες έχουν ήδη αναλάβει νομικά τη δέσμευση, να αναγκαστούν ενδεχομένω να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Και όπως είπα, μία ή δύο ίσως να υποβάλουν και αίτηση ένταξη στην Ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια. Δεύτερο, όταν ε, ήμουν επικεφαλής της ειδική Επιτροπής για την Δημοσιονομική Κρίση και με την Περβάνς Μπερές είχαμε κοιτάξει και τους οίκου αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν επιθυμητό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που να μην εξαρτάται από αμερικανική επιρροή. Και σύμφωνα με τις ιδέες που είχαμε ε, αναπτύξει τότε θα πρέπει να είναι ιδιωτικός οργανισμός, όχι δημόσιος, ε, όμως ε, να λάβει και επένδυση από δημόσιο χρήμα και να μπορέσει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο, το business model και να εξαρτάται και από τους επενδυτές και όχι μόνο από τις εκδόσεις ε, ε, εγώ το προωθώ το ε, σχέδιο αυτό, το έχω κάνει προσωπική μου υπόθεση και ψάχνω να βρω επενδυτές οι οποίοι να συμμετάσχουν. Γιατί ως την ώρα το διάβημα αυτό δεν ήταν επιτυχές. Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι ένας αριθμός τέτοιων οργανισμών έχουν αρχίσει να λειτουργούν. Και ένας από αυτούς με 200 μέλη προσωπικό και λειτουργεί ήδη σε 6 χώρες έχει γίνει μάλιστα αποδεκτός και από επιχειρήσεις αλλά και θεσμούς όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτοί οι άνθρωποι μου λένε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να μην τους θεωρεί ισότιμους με, τα, με τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης της πιστολεπτικής ικανότητας, standard pools κτλ. Απάντηση για την πρώτη σας ερώτηση. Η ζώνη έχει ενισχυθεί. Παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε εμείς να δούμε και ταχύτερους ρυθμούς. Έχει γίνει πάντως πρόοδος και ιδίως αν εξετάσει κανείς, αν λάβει δηλαδή ως αφιτηρία την αρχή της κρίσης. Η διαδικασία λοιπόν αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως έχει προχωρήσει επαρκώς, ώστε να μπορώ να αντιστρέψω το ερώτημά σας. Δηλαδή, έχουμε και πρόσφατα εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και αυτές το επιβεβαιώνουν. Η κύρια έμφαση δεν είναι πλέον στο ερώτημα αν η Ευρωζώνη είναι ικανή να διευρυνθεί, αλλά εάν κάποια χώρα μέλος είναι ικανή να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Αναμένουμε λοιπόν χώρες μέλη της Ένωσης που δεν έχουν περιλάβει στις ε, συνθήκες τους ρήτρα opt-out, αναμένουμε να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Αυτό, που θα, αυτό θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες. Την προθυμία τους και την ικανότητά τους. Η ικανότητά τους είναι μια διαδικασία, υπάρχει διαδικασία δηλαδή με μια μεγάλη διαφορά ε, ως προς το παρελθόν. Οι χώρες αυτές πρέπει να είναι ε, να αντιληφθούν δηλαδή ότι τώρα εντάσσονται και σε τραπεζική ένωση. Επομένως θα υπάρχει μια διαδικασία όπου η ένταξή τους στην Ευρωζώνη, οι χώρες αυτές εφόσον ενταχθούν, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι και οι τράπεζές τους θα κληθούν να ενισχύσουν την Τραπεζική Ένωση και όχι να προκαλέσουν νέες ρογμές και νέες ε, ευαισθησίες αυτή είναι η, η απάντηση στην πρώτη σα ερώτηση. Είμαστε σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Όταν διαρωτώμεθα τότε έχει νόημα η διεύρυνση αυτή. Μήπως θα αποδυναμώσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά ε, πράγματα έχουν αλλάξει όμως από τότε. Και όπως είπα, πρέπει να αλλάξουμε ώστε να μπορέσει και η Ένωση να γίνει ισχυρότερη. Ξεκινώντας από τη σημερινή εφετηρία, κρίνω ότι είμαστε αρκετά ισχυροί, ω Ευρωζώνη δηλαδή τώρα, για να απορροφήσουμε και νέα μέλη. Το δεύτερο τώρα για τους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας. Μπορούμε να συζητήσουμε εάν η οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας είναι τέλη ή όχι. Όταν επικεφαλής της FSB και δίνοντας την πρώτη απάντηση στην πρώτη ε, δημοσιονομική κρίση του 2008, ο ρόλος που είχαν παίξει οι οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας, ο ρόλος τους δεν ήταν, πώς να πω, διόλου αξιοσύστατος, διόλου αξιέπαινος, ας πούμε έτσι. Και είχα πει τότε ότι θα πρέπει να μπορούμε να λειτουργήσουμε και χωρίς αυτούς. Γεγονός πάντως είναι ότι έκτοτε φάνηκε ότι είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν με κάτι. Και όταν ε, μιλώ για αντικατάσταση εννοώ κάτι που να του αντικαταστήσει και που θα ε, απολαμβάνει όμως το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης από τους βασικούς θεσμικούς επενδυτές, δηλαδή στα αξιοδοτικά ταμεία και όλους τους άλλους βασικούς φορείς στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Διότι αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των οίκων αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητας, οι οποίοι οίκοι να χάσουν την εμπιστοσύνη αυτή, διότι είχαν δώσει συμβουλές στους επενδυτές να αγοράσουν προϊόντα τα οποία πραγματικά δεν άξιζαν τον κόπο να αγοραστούν. Είναι πολύ δύσκολο ωστόσο να... αυτό το πω ε, ε, Εάν ο οργανισμό αυτό είναι ιδιωτικό, ασφαλώς θα χαίρει μεγάλη εμπιστοσύνη παρά εάν είναι δημόσιο. Από την άλλη μεριά όμως είναι δύσκολο να μπει κανεί στην αγορά αυτή όταν είναι απ' έξω. Ασφαλώς και θα θέλαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας μπορούμε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ξέρω για αυτόν τον οργανισμό που λέτε, που τον αποκαλείτε SCOPE. Θέλουμε όμως Έχουμε βέβαια του οίκου πιστοληπτική ικανότητα. έχουμε όμω και άλλε αξιολογήσει, γιατί και οι κεντρικέ τράπεζε έχουν τι δικέ του αξιολογήσει, υπάρχουν και εσωτερικέ αξιολογήσει πιστοληπτική ικανότητα. Αλλά ασφαλώ είμαστε ανοιχτοί απέναντι στο ενδεχόμενο, τη δυνατότητα διεύρυνσης όσο γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Στέφαν Γκέρολτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε εδώ κοιτά. Αναφερθήκατε σε Βορρά και Νότο. Που ενώνει το ευρώ. Αλλά οικονομικά είναι πολύ διχασμένο. Για τη συνοχή της Ευρωζώνης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε επιλέξει χαμηλό επίπεδο επιτοκίων. Με συνέπεια όμως για το... τα κράτη που έχουν χρέη όπως άλλωστε είχε προβλεφθεί. Αλλά για, τους, ε, για ποιον έχει αποτομίευση, τι συνέπειες θα έχει αυτό. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διακοπή του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα εργαλεία ή βαλβίδες προσαρμογής για να γίνεται αυτή πιο πρόσκοπτα. Κύριε Ντράγκη, εάν μπορούσατε εσείς να εκφράσετε την ευχή για ένα ακόμα εργαλείο στην εργαλειοθήκη σας, στην και της Ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποιο θα ζητούσατε. Ευχαριστώ. Ντράγκη. Ευχαριστώ. Χαμηλό και αρνητικό ακόμη επιτόκιο που έχουμε. Το χαμηλό αυτό επιτόκιο δεν έχει σαν στόχο τη διατήρηση της συνοχής τη Ευρωζώνης. Ε, ο στόχος ήταν περισσότερο αυτό που θα ονομάζαμε αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης. Ε, πάνω απ' όλα ωστόσο ήταν η σταθερότητα των τιμών. Γιατί τα τελευταία χρόνια και σε κάποιο χρονικό σημείο της κρίσης κατέστη σαφές ότι μπορούσε αυτό το εργαλείο να φέρει πολύ πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως άλλωστε αποδείχθηκε από, τη θετική, το θετικό αντίκτυπο των αρνητικών επιτοκίων ως ε, παράγοντα μοχλό για την οικονομία αλλά και για την υπέρβαση της χρηματοπιστωτικής ε, ε, του χρηματοπιστωτικού κατακαιρματισμού. Τώρα, συνέπειες για την αποταμίευση. Να το κοιτάξουμε. Το αρνητικό είναι μόνο μια πολύ βράχη πρόθεσμη πολιτική επιτοκίων. Αλλά είναι αμφίβολο το αν όντω συμφέρουν η ε, αποτεμιεύσει αυτό το βράχη πρόθεσμο ε, διάστημα ε, γιατί η αποταμίευση φερειπίν για τις επιχειρήσεις αποταμίευση μιλάω, καταθέσεις μιλάω, δεν είναι μηδενικές, ε, μηδενικά τα επιτόκια των ε, καταθέσεων απαραίτητα και μάλιστα δεν γίνονται απαραίτητα οι επενδύσεις σε πρόθεσμο στοιχείο όπως είναι ε, το ταμιευτήριο, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αλλά σε άλλες μορφές επενδύσεων. Τώρα για να κρυφεί η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου θα πρέπει κανείς να κοιτάξει ευρύτερα ζητήματα όπως είναι πιο συμφέρον η αποταμίευση σε μια ισχυρή οικονομία με, μείωση της ανεργίας να γίνεται, να γίνεται η αποταμίευση εκεί είναι καλύτερο για, τον, ε, ε, ε, για την αποταμίευση αυτό ή θα ήταν καλύτερο με υψηλότερα επιτόκια σε μια πιο πτυτική οικονομία με λιγότερες θέσεις εργασίας, με χαμηλότερους μισθούς κτλ. Άρα λοιπόν να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση, νομίζω η απάντηση είναι ότι το πολύ χαμηλό ιανητικό επιτόκιο έχει διαδραματίσει πολύ θετικό ρόλο για την νομισματική πολιτική και με βάση βέβαια τόσο ορίζει η εντολή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώνεται το κομμάτι του διαλόγου μέσα ως, πρόεδρο, διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, τώρα περνάμε στο κομμάτι που αφορά την ε, διαχείριση του συστημικού κινδύνου με εσάς ως πρόεδρο της Επιτροπής ε, Συστημικού Κινδύνου και ξαναδίνω το λόγο στον πρόεδρο Ντράκη. Ας πιω λίγο νεράκι πρώτα. Μην το ξεχάσετε αυτό, λέει ο κύριο Φέρπες. Όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Πολύ γενναιόδωρο. Honorable members of the Economic and Monetary Κυρίε και κύριοι, μέλη της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος τώρα της Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου και όπως είπα, τελευταία συνεδρία στην τρέχουσα θητεία και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας μιλήσω για την πρόοδο που έχουμε επιτύχει στην μακροπροληπτική ε, πολιτική με τις ε, προσεγγίσεις που ε, θα δημοσιευθούν σήμερα και να συστήσουμε και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε λοιπόν σημαντική επιτυχία γιατί αποτελούμε μια ε, ένα κέντρο για την εξέταση των δυσκολιών, αλλά ταυτόχρονα και ένα κέντρο που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον με την ε, εμπειρία που ανταλλάσσουμε και την χρήση των μακροπροληπτικών εργαλείων, αλλά ταυτόχρονα και δράσεις μακροπροληπτικές μπορούμε να αναλάβουμε με μια νέα όθηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρήση αυτών των εργαλείων ήπη ε, ενδοτικού δικαίου, όπως ονομάζονται, που είναι οι συστάσεις για την καθοδήγηση των δράσεων. Στις αρχές λοιπόν του, της περίοδου αυτής της βουλευτικής εξασφαλίστηκε για τις αρχές μακροπολιτικής καθοδήγησης η πρόσβαση στα εργαλεία που απαιτούνται ως ρυθμιστική απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση και κατά τη συνεδριάση μας συζητήσαμε πώς οι αρχές αξιοποιούν τα εργαλεία αυτά για να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους και σε απάντηση των συστάσεων του, ε, της ρυθμιστικής αρχής ε, με τις συστάσεις και τις προειδοποίησεις για τα σημεία τα πιο ευάλωτα για τον τομέα των ε, ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι αρχές λοιπόν, μακροπροκριτικές αρχές έχουν την ε, βούληση να χρησιμοποιήσουν τα μέσα, τα εργαλεία πολιτικής που υπάρχουν και τα δραστηριοποιούν κατά τρόπο στοχευμένο, επί παραδείγματι. Το buffer συστημικού κινδύνου, το μαξιλαράκι συστημικού κινδύνου χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικοί κίνδυνοι για 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την ε, Νορβηγία. Υπάρχουν λοιπόν ε, διαφορές με ένα ε, απόθεμα τέτοιο που ποικίλει από το 0,5% στο 2% και ακόμη πέντε χώρες έχουν ένα θετικό ποσοστό για το επόμενο 12 μήνο με 0,25% έως 2,5%. Επιπλέον δε στην πλειονότητα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μακροπροληπτικές αρχές έχουν αξιοποιήσει εργαλεία με βάση το δανεισμό που είναι διαθέσιμα στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για να εξασφαλίσουν υγιείς συνθήκες δανεισμού και να περιορίσουν τον κίνδυνο ε, υπερβολικού δανεισμού των οικοκυριών. Και έτσι φτάνω στην έκθεση του ESRB για την ε, μακροπροληπτική προσέγγιση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Επιτρέψτε μου λοιπόν ε, σύντομα να συνοψίσω τις κύριες ε, ανησυχίες που προκύπτουν σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ε, όταν λοιπόν υπάρχουν πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και συσσωρεύονται αυτά μπορεί να αποτελέσουν ε, πρόβλημα εάν επηρεάζουν σημαντικό κομμάτι του χρηματοπιστωτικού συστήματο, εάν περιορίζουν την ανθεκτικότητά του στου κλειδονισμού, εάν παρεμποδίζουν την κύρια λειτουργία του ε, που είναι η διευκόλυνση ε, των οικονομικών συναλλαγών. Δεδομένης λοιπόν τη εντολή και του προηγούμενου ρόλου στην επίλυση με εξυπηρετούμενων, θεμάτων σχετικών με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ECRB, ζητήθηκε από το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. το να αναπτύξει προσεγγίσεις μακροπροληπτικές για την αποτροπή της εμφάνισης ε, συστημικού τύπου ή συστημικής έκτασης ε, προβλημάτων σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι δημοσιεύουμε σήμερα την έκθεση όπου συμπεραίνουμε πως ήδη υπάρχουν επαρκή εργαλεία για την αντιμετώπιση των ευάλωτων σημείων. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τις τελευταίες αλλαγές στο μακροπροληπτικό ε, πλαίσιο για το απόθεμα ασφαλείας που απαιτείται ε, ότι θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την ευελιξία του συστημικού αυτού αποθέματος και θα εξοπλίσει τις μακροπροληπτικές αρχές με στοχευμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση θυλάκων ε, ε, ευάλωτων ή συγκεκριμένων τομέων της αγοράς ή συγκεκριμένων ομάδων ε, δανειοληπτών. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε εντοπίσει τομείς όπου χρειάζεται περισσότερη δουλειά και θα ήθελα να τους περιγράψω αυτούς τους τομείς, κυρίως σε σχέση με τα μέτρα που αφορούν τον δανειολήπτη. Με λίγα λόγια. Ανώτατο όριο στο δάνειο με βάση την αξία ή στο δάνειο με βάση το εισόδημα ε, είναι ελάχιστες προδιαγραφές που μπορούν να επιβληθούν. Δηλαδή ο δανειολήπτης ε, δεν μπορεί να υπερχρεωθεί και άρα να καταστεί πιο ευάλωτο σε οικονομικούς, οικονομικούς ε, κλειδονισμούς. Έτσι λοιπόν τα μέτρα αυτά ταυτόχρονα ενισχύουν και την ανθεκτικότητα των τραπεζών περιορίζοντας την ποσότητα, τη μάζα δανείου που μπορεί να έχει να κάνει με τις εγγύησεις με το εισόδημα του δανειολήπτη και έτσι μπορούν να περιορίσουν τον την ε, ε, υπερβολική αύξηση των πιστώσεων. Με τον τρόπο αυτό συγκρατείται ο κίνδυνος σε προώρο στάδιο. Όπως ήδη έχω αναφέρει τα μέτρα αυτά που στοχεύουν τον διαλυολήπτη, ήδη χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε κράτη-μέλη ε, στο δανεισμό προς τα νοικοκυριά και η CRB θεωρεί ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις μακροπροληπτικές αρχές, πράγμα το οποίο δεν ισχύει αυτή τη στιγμή επιπλέον. Δεδομένων και των ε, πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν τα εργαλεία αυτά, τα μέτρα αυτά. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλους δανειολήπτες, όχι μόνο στα νοικοκυρά δηλαδή, μη χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα ε, εταιρείε. Και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω. Βέβαια, ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο ένα τέτοιο επιχείρημα και γιατί είναι εταιρεογενή πολύ ο τομέα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ω προ το μέγεθο, ε, τον τομέα την ε, ε, ηλικία τους, τη διάρκεια δηλαδή παρουσία τους στην αγορά και των δανείων που μπορεί να τους χορηγούνται. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ποια είναι τα ευάλωτα στοιχεία και ποιοι είναι οι διαρθρωτικοί παράγοντες που μπορεί να χαρακτηρίζουν ε, πιθανά προβλήματα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως είναι η ανεπάρκεια σε νομικό και δικαστικό πλαίσιο ή στην διαχείριση των τραπεζών, που είναι έξω βέβαια από το προληπτικό τομέα. Ταυτόχρονα όμως προσδιορίζονται και οι παράγοντες, οι συνθήκες μέσα στις οποίες ε, λειτουργεί η μακροπροληπτική πολιτική. Άρα πρέπει να καλυφθούν τα προβλήματα, τα κενά σε νομικό και δικαστικό επίπεδο που ήδη υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ τώρα στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, δεδομένου ότι η πιστοτική διαμεσολάβηση ασκείται από μη τραπεζικούς φορείς, χρηματοπιστωτικού φορείς, η Ευρώπη θα πρέπει να εξοπλίσει τις μακροπροληπτικές αρχές με τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου, ε, εάν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, να τους μεταφέρει έξω του τραπεζικού τομέα ή να τους προλάβει. Έτσι λοιπόν στην Επιτροπή αυτή συχνά έχω συζητήσει τη στρατηγική του ESR, στην Επιτροπή σας έχω συχνά συζητήσει τη στρατηγική του ESRB και τις προτεραιότητες μας για την επέκταση της ε, μακροπροληπτικής ε, πολιτικής επέμβασης πέραν των, του τραπεζικού τομέα και κατά τις συνεδριάσεις μας συζητήσαμε τις προτάσεις μας για την αναθεώρηση του ΕΜΙΡ, του κανονισμού δηλαδή για τις υποδομές τραπεζών ε, ε, ευρωπαϊκής αγοράς. Ταυτόχρονα την πρώτη τελευταία φορά που συναντηθήκαμε τόνισα τα στοιχεία εργαλείων που μπορούμε να προτείνουμε για τον ασφαλιστικό τομέα με την ε, αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητα και κινδύνων που σχετίζονται με τη μόχλευση σε ορισμένε περιπτώσει επενδυτικών ταμείων. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να πω ότι δυστυχώ εδώ ε, δεν σημειώθηκε σημαντική η επαρκή πρόοδο ω προ την ενσωμάτωση των μακροπροληπτικών εργαλείων στον τομέα των μη τραπεζικών στο νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια άλλη πρόκληση μπροστά μα σχετίζεται με την παρακολούθηση, με την επιτήρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας λεπτομερή αλλά και διάχυτα ε, στοιχεία συναλλαγών, για να έχουμε δηλαδή μια πλήρη εικόνα, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε τις αγορές και να συνδυάσουμε τα, δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε από τις αγορές, με βάση τα εργαλεία ή τα συναλλάγματα, τα ανταλλάγματα που προσφέρονται. Η εμπειρία μας στην ανάλυση των ε, παραγόγων δεδομένων που μας εξασφαλίζουν ε, το ΕΜΙΡ ε, δίνει πολύ μεγάλη σημασία, αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη σημασία της μεγαλύτερης τυποποίησης των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο μάλιστα ή δυνατόν, αλλά και τη βελτίωση της ανάλυσης των αναλυτικών εργαλείων. Θα ήθελα ολοκληρώνοντα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της για την εξαιρετική εξαιρετική συνεργασία τα τελευταία χρόνια και την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων όχι μόνο εδώ αλλά και στις και των θυρών όπως προβλέπετε, συνεδριάσεις μας. Ιδιαίτερα ε, ικανοποίηση αισθάνομαι για τα δύο θέματα στο οποία έχετε δώσει ιδιαίτερη προσοχή που έχει να κάνει με τις ε, συνέπειες της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις, ε, το πρότυπο υπαριθμών 9 για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Έτσι λοιπόν έχουμε προχωρήσει και εμείς σε δημοσιεύσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς. Ελπίζω ότι θα μπορέσω σε μελλοντική συνεδρίαση να σας ενημερώσω για το περαιτέρω έργο μας που συνεχίζεται. Θα μελετήσουμε βεβαίως και τις χρηματοπιστωτικές συνέπειες των ε, ε, του προτύπου παριθμών 17 από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα σε σχέση με τις ασφαλιστικές συμβάσεις δηλαδή. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την παρουσία της κυρίας Μπερβάνς Μπέρες και του κυρίου Μπούρχατ ε, ε, Μπάλτς εκ μέρους της Επιτροπής σας σε μία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ECRB. Ελπίζω ότι αυτό διευκόλυνε το έργο σας και την επισκόπηση των βασικών, του βασικού μας κανονισμού λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξάλλου ευχαριστούμε που υπενθυμίσατε και τις συνεργασίες στις καταστατικές μας ε, ε, συνεδριάσεις. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω την σημασία των όσων είπατε. σχετικά με την επέκταση του φάσματος της μακροπροληπτικής ε, πολιτικής και πέραν των τραπεζών και έχουμε πράγματι σημειώσει πρόοδο στον τομέα αυτό. Σημαντικό για όλο μας το έργο και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, να προσπαθήσουμε να είμαστε συντομότεροι και συντομότερες, διότι έχει και αεροπλάνο να προλάβει ο πρόεδρος Ντράγκη. Πρώτος ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε. Έχω να θίξω ένα θέμα που βλέπω συστημικό κίνδυνο. Δηλαδή τι ανταλλαγές swap line που έχουμε με την ε, Τράπεζα της Αγγλίας. Σε περίπτωση σκληρού Brexit, τι θα γίνει με το swap line, τι, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ποιες είναι οι παράμετροι, προσαρμόζονται, έχει μειωθεί ο όγκος προτίθεστε να μειώσετε τον όγκο εν ώψη του Brexit και αν ναι σε ποιο βαθμό, με ποιες συνθήκες και βεβαίως και συνεργασία με τις εθνικές τράπεζες οι οποίες ε, σε αρνητική περίπτωση θα πρέπει να ε, αναπληρώσουν τα κενά. Και βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και προβλήματα με το Euro Clearing. Υπάρχουν λαμβάνονται μέτρα ποια είναι τα νομικά μέτρα ιδίω για το Euroclearing και ιδίω για το LCH που είναι ένας, κυρίως ένας από τους οίκους clearing, συμψηφισμού δηλαδή, που ε, ενδέχεται να πληγούν από αυτό. Ο πρόεδρος Τράγκη. Δύσκολο να συζητήσω όλα αυτά τα θέματα τώρα. Αφενός, τουλάχιστον το τελευταίο μέρος της ερωτήσεως σας για το Brexit. Εμείς δεν συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να, δύσκολο να συζητήσουμε ενδεχόμενα. Μπορώ να επαναλάβω αυτό που είπα πριν. Έχουμε προετοιμάσει το έδαφος. Μαζί με την Τράπεζα της Αγγλίας έχουμε εντοπίσει τομείς που είναι ευάλωτοι και έχουμε δει τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει προσφέρει επαρκή χρόνο για να αντιμετωπιστούν τα διάφορα σενάρια. Δίνονται δηλαδή, ε, δίνεται επαρκής χρόνος για να ληφθούν μετριαστικές δράσεις. Αν δεν, υπάρξει, δεν υπήρξαν μάλλον καθόλου κινήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό σημαίνει ότι όλοι είναι παγωμένοι και αναμένουν, αναμένουν να δουν τι θα γίνει. Και μετά θα αποφασίσουν. Το ίδιο ισχύει για την swap line. Δεν μπορώ να συζητήσω για ενδεχόμενα, δηλαδή πώς, πότε και εάν. Είναι η μοναδική σου που έχουμε. Δεν... Πάντως, είναι καλός συνομιλητής η Τράπεζα της Αγγλίας για swap για ανταλλαγές δηλαδή. Αυτό θα πρέπει να είναι επαρκές για να καθησυχάσουμε όλους ενδιαφερομένους ότι και τα δύο μέρη ναι, αλλά αυτοί που φέρουν τους κινδύνους γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Αυτοί γνωρίζουν ενήμεροι για τις λεπτομέρειες του Σόπλαιν. Ναι, όλοι όσοι φέρουν τους κινδύνους, δηλαδή όλα τα μέλη του Συμβουλίου γνωρίζουν τα σχετικά, αλλά ξαναλέω δεν είναι η μόνη Σόπλαιν που έχουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο κίνδυνο άνευ προηγουμένου που ε, διατρέχουμε. Καλωσορίζω τον νέο μέλος, την κυρία Βίντερ δηλαδή. Καλώς ήρθατε στην ε, ε, ε, Επιτροπή Οικονομικών. Ευχαριστώ. Ερώτηση, αλλά στη γερμανική γλώσσα. Αξιότιμη κύριε Τράγκη, όπως μόλις είπε ο πρόεδρος, είμαι νέο μέλος της Επιτροπής Οικονομικών. Δεν έχω τη δυνατότητα να συγκρίνω με τους προηγουμένους διαλόγους, αλλά μετά από αυτές τις δυόμιση ώρες που ε, παρακολούθησα τη συζήτηση εδώ. Ε, θεωρώ πραγματικά και εγώ ότι είναι ιδιαίτερα ε, σημαντική η ενημέρωση βεβαίως και για όσα θέλουμε να μεταφέρουμε και εμείς στους ψηφοφόρους μας. Ασφαλώς και κινούμεθα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού εδώ, αλλά ως βουλευτής είμαι υπεύθυνη και απέναντι στους ψηφοφόρους μου και πρέπει να τους μεταφέρω πληροφορίες. Έχω τώρα δύο πράγματα να ερωτήσω. Αφενός μια γενική ερώτηση για το προγνωστικό ανάπτυξης. Δηλώσατε προηγουμένως ότι οι προγνώσεις για την ανάπτυξη έχουν μειωθεί. Η ερώτησή μου από την άποψη του Συμβουλίου θεωρείτε ότι κινούμεθα μέσα σε ένα ε, κύκλο συγκυρίας ή θεωρείτε ότι βρισκόμαστε εκτός κύκλου. Δεν θέλω κι εγώ να θέσω τώρα ως δεύτερη ερώτηση, ερώτηση για, την, για το Brexit, όπως για παράδειγμα τιμωρητικούς δασμούς, που επίσης και αυτή η συζήτηση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις προγνώσεις ε, της ανάπτυξης. Δεύτερη ερώτηση πάντως, κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα το κοινό στη Γερμανία. Πρόκειται για φήμες ή και συζητήσεις και στα μέσα για ενδεχόμενη συγχώνευση δύο τραπεζών, της Deutsche Bank και της Commerzbank. Δεν σας καλώ τώρα να τοποθετηθείτε απέναντι σε μια συγκεκριμένη συγχώνευση, αλλά θέλω να σας ερωτήσω μια συγχώνευση που υποτίθεται ότι θα εξασφαλίσει την κερδοφορία, πάντοτε συνεπάγεται και τον κίνδυνο της απώλειας θέσεων απασχόλησης. Από την άλλη μεριά μεγαλώνει η τράπεζα. Μήπως μπαίνουμε σε ένα κίνδυνο τότε too big to fail, κάτι το οποίο εν τέλει θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους και οι φορολογούμενοι τουλάχιστον στην Γερμανία ανησυχούν πάρα πολύ για το ενδεχόμενο αυτό. Πώς το βλέπει αυτό το ε, Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. θεωρεί ότι είναι προτιμότερη μία εκδοχή, δηλαδή τη συγχώνευση, ή οι άλλοι, δηλαδή να παραμείνουν δραστήριε και οι δύο τράπεζε. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση για τον κύκλο ανάπτυξης. Όλα αυτά τα στοιχεία, ασφαλώς, το 2017 ήταν ένα εξαιρετικό έτος ό,τι αφορά την ανάπτυξη και αυτή οφειλόταν ιδίω στην εξωτερική ζήτηση, δηλαδή στις εξαγωγές, οι οποίες τα πήγαν πολύ καλά. Εν μέρη λοιπόν αυτή η πτώση είναι ίσως αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή μια προσγείωση σε μια τροχιά χαμηλότερη, όμως κοντά στο δυναμικό. Αυτό τι γίνεται τώρα πέραν αυτού. Αυτό θα είναι ένα μείγμα εξειδικευμένων παραγόντων, εξειδικευμένων αναχώρα δηλαδή, ή και ενδεχομένως γεγονότων και γεωπολιτικών γεγονότων. η ζήτηση από τον υπόλοιπο κόσμο έχει μειωθεί και αυτό εν μέρη οφείλεται και στην απειλή προστατευτισμού που νομίζω το είπα και πριν αυτό εάν γνωρίζαμε ότι είναι κυκλικός ο χαρακτήρας αυτός θα εξαφανιζόταν ένα μεγάλο μέρο τη αβεβαιότητα. Βέβαια, υπάρχει και μεγάλη συζήτηση και μακρά συζήτηση περί Brexit, η οποία θίγει την εμπιστοσύνη και εντό τη ζώνη ευρώ. Και βέβαια, έχουμε και πολιτικέ εξέλιξει σε πολλέ χώρε και τη ευρωζώνη, που και αυτέ ε, μειώνουν την, ε, ή τέλο πάντων ε, θίγουν την εμπιστοσύνη και μειώνουν την ε, ανάπτυξη. Έχουμε τώρα και Έχουμε τώρα και την ανάπτυξη στην Κίνα που μειώνεται επίσης. Έχουμε την μείωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την μείωση της παραγωγής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία. Πρόκειται δηλαδή για ένα συνδυασμό γεγονότων που όλα αυτά συνδυάζονται και έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θεώρησε ότι ναι μειώνεται τώρα η ανάπτυξη, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι η επιμονή των αποτελεσμάτων αυτών και ιδίω αυτών που δεν είναι εφάπαξ μόνο. Η αβεβαιότητα, για παράδειγμα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Εάν επιμείνει, τότε αυτό το slowdown θα είναι μακρύτερο. Για την ώρα, η πιθανότητα ύφεση για την Ευρωζώνη είναι χαμηλή για το σύνολο της Ευρωζώνης. Εξάλλου όμως βλέπουμε ότι η υπόλοιπη οικονομία στο σύνολο της ε, Ευρωζώνης βελτιώνεται. Η αγορά εργασίας, για παράδειγμα, ε, είναι στα ωριά της. Κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν όρια στην ανάπτυξή τους λόγω έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και γι' αυτό θεωρούμε ότι συγκρίνουμε προς τον στόχο μας. Αν όμως η επιβράδυνση αυτή συνεχίσει, τότε ίσως η ανάκαμψη να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Θα δούμε τον Μάρτιο τα πράγματα αυτά όταν θα δημοσιεύσουμε τις προβλέψεις του Μαρτίου για την Ευρωζώνη. Τώρα για το δεύτερο δεν μπορώ να σχολιάσω για επιμέρους ε, ιδρύματα. Ναι, κάπως ξεπερνώ τον χρόνο μου. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Ε, εάν κάποια ιδρύματα μεγαλώνουν ή αν έχετε ήδη μεγάλα, υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενδεχόμενο κινδύνου too big to fail. Πρώτα-πρώτα ε, διασύνδεση. Τι να γίνει σε περίπτωση ε, εξυγίανσης, εποπτεία. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αυτός. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα τραπεζικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλα ώστε να μην μπορεί να επιτραπεί να πτωχεύσουν. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να τίνουμε προς ένα βέλτιστο μέγεθος και κλίμακα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Θα επανέλθω στο θέμα των κόκκινων δανείων, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ανησυχία σε εκατομμύρια Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν φτωχοποιηθεί από την πολιτική των μνημονίων τα τελευταία 8 χρόνια. Και φυσικά ρωτούν οι ίδιοι τελικά θα υπάρξει ένα σχέδιο διάσωσης των φτωχών δανειοληπτών. Γιατί διασώθηκαν οι ελληνικές τράπεζες και αυτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και ρωτούν επίσης μπορεί να δημιουργηθεί ταμείο σωτηρίας δανειοληπτών με κρατικά χρήματα. Υπάρχει και η άποψη ένα ειδικό όχημα διάσωσης των δανειοληπτών από την ε, Τράπεζα της Ελλάδος. Ρωτούν επίσης οι δανειολήπτες. Καλά, είναι λογικό να πολιθούν τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια στα funds σε μια τιμή 8-10% και να μην μπορούν στην ίδια τιμή να τα αγοράσουν οι δανειολήπτες. Είναι απλά πράγματα κύριε Ντράγκη και μάλιστα έχουμε και ευρωεκλογέ και οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ένας ε, δανειολήπτης με ένα δάνειο 100.000 ευρώ στεγαστικό λέει αυτό το δάνειο μπορεί να το αγοράσει το φαντ με 10.000 ευρώ. Γιατί να μην μπορεί να το αγοράσει αυτό το δάνειο ο ίδιος ο δανειολήπτης σε αυτό το ποσό. Γιατί να μην μπορεί να αγοράσει αυτό το δάνειο ένα κρατικό όχημα, μια κρατική εταιρεία και εν συνεχεία ο δανειολήπτης να εξοφλήσει αυτά τα ποσά. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις. Προηγουμένως απαντήσατε αόριστα και γενικά και θα ήθελα πολύ πιο συγκεκριμένα να δώσετε μια απάντηση. Μας παρακολουθούν οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή ανησυχούν ότι θα χάσουν τα σπίτια τους στους πληστηριασμούς και θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα αυτό. Εσείς ως Κεντρική Τράπεζα βλέπετε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα κρατικό σχήμα το οποίο θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, θα διασώσει τους δανειολήπτες και στην πορεία οι δανειολήπτες θα μπορούν να αγοράσουν τα δάνειά τους από αυτή την κρατική εταιρεία. Ευχαριστώ απάντηση. Είπα και πριν, τώρα συζητιέται αυτό στην Αθήνα, οπότε δεν μπορώ να το συζητήσω εδώ τώρα. Τι μπορεί να πει κανείς. Είναι ότι βέβαια πάντα μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα ειδικό όχημα από το κράτος, να αγοράσει και να δούμε σε ποια τιμή. Αλλά το ζήτημα εδώ που προκύπτει είναι το φαντ που αγοράζει αυτά τα δάνεια και άρα βοηθάει τους φτωχού δανειολήπτες μεταξύ των ε, πιστωτών μπορεί να δημιουργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε κατά υπέρ κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιστεύει ότι το κοινωνικό σκέλος του προβλήματος, γιατί είπα και πριν, υπάρχουν εδώ δύο σκέλη. Υπάρχουν οι πραγματικά φτωχοί και υπάρχουν και οι στρατηγικά φτωχοί. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι διαφορετική. Για τους φτωχούς δανειολήπτες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν και οι κοινωνικές τους ε, αδυναμίες, τα κοινωνικά τους προβλήματα, χωρίς όμως να καταστραφεί το σύστημα. Τώρα η αποστολή βρίσκεται στην Ελλάδα και το συζητάει. Πρέπει να συμμορφωνόμαστε όμως και με τους κανόνες. Ένα λεπτό έχω, δεν το έχω ολοκληρώσει, λέει ο κ. Μαριάς. Λοιπόν. Το δάνειο 100.000 ευρώ το αγοράζει το φαντ 10.000 ευρώ. Γιατί να μην αγοραστεί σε αυτή την τιμή το δάνειο από τον ίδιο το δανειολήπτη. Και επειδή δεν μπορεί ο ίδιος ο δανειολήπτης να το κάνει, να το αγοράσει αυτό ένα κρατικό ίδρυμα. Πρέπει να βρούμε μια ρύθμιση στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Βρήκαμε τέτοιες ρυθμίσεις παλαιότερα για τις τράπεζες. Γιατί να μην βρεθεί μια ρύθμιση τέτοια για τους δανειολήπτες. Thank you. Μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική κυβέρνηση θα το αποφασίσει, όχι εμείς. Πρόεδρος Ραμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Καλκέρη, Πρόεδρε Δράγκη. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή αυτή και πάλι. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια και το εξαιρετικό έργο που έχετε επιτελέσει. Για να βγούμε από την οικονομική κρίση. Ε, πολύ μου άρεσε η συζήτηση ανάμεσα σε εσά και τον κύριο Λάμπριτ ε, για του δεσμευτικού κανόνε όσον αφορά τη σύγκληση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε όταν δεν είναι δεσμευτικοί κανόνε και είπατε επίση ότι όταν είναι το δημόσιο χρέος ιδιαίτερα υψηλό, οι χώρες χάνουν σε κυριαρχία. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε λίγο για την περίπτωση αυτή του υψηλού χρέους. Έπειτα, έχουμε δει αποκλίσεις ανάμεσα στις μεγάλες χώρες στην Ευρωζώνη. Έχουμε τη Γερμανία που βελτιώνει την κατάσταση από 80-60%. Άλλες χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αυξάνουν το έπτους και τη σχέση με το χρέος. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τη διαχωριστική γραμμή. Όταν έχουμε τράπεζες μιας χώρας που έχουν υπερβολικά πολλά ε, δάνεια, δεν ξέρω εσείς την εξέλιξη πώς τη βλέπετε τα επόμενα χρόνια. Έπειτα όσον αφορά την αγορά ομολόγων, οι εγγύσει για τις τράπεζες παραμένουν ίδιες. Δεν γίνεται κούρεμα. Είδαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο ότι ελοχεύουν κίνδυνοι. Οπότε οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές θα πρότειναν κούρεμα για το κρατικό χρέος ή όχι, για να πετύχουμε τη σταθερότητα. Ευχαριστώ. Είναι βέβαια δύσκολο να πει κανείς πότε είναι ιδιαίτερα υψηλό. Υπάρχει βέβαια νέα θεωρία, διάφορες θεωρίες, χωρίς να μπούμε στις λεπτομέρειες, θα επικεντρωνόμουν μόνο σε μία πτυχή. Ο τρόπος που μειώνονται τα χρέη, με το παράδειγμα που δώσατε κι εσείς στην Ευρωζώνη, είναι κυρίως όταν πριν η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Είναι πολύ βασική για να μειωθεί η σχέση χρέους ΑΕΠ. Είναι προφανές αυτό. Οπότε, όλες οι χώρες στην Ευρωζώνη, δείτε τα τελευταία δέκα χρόνια, ακολούθησαν μια δημοσιονομική πολιτική που ήταν σε λογικά πλαίσια μισό, ένα εκατό, παραπάνω, παρακάτω. Πάντως γενικά ήταν λογική. Αυτό το ζωτική σημασία και παραμένει είναι μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν ε, στην ανάπτυξη να επανέλθει την οικονομική μεγένθηση και στο παράδειγμα που δίνεται για τη Γερμανία. Αυτό ακριβώς έκανε η Γερμανία στις αρχές του 2000 και άλλες χώρες το έκαναν το ίδιο. Και γι' αυτό μειώνεται το χρέος. Έτσι, όχι επειδή υπήρξαν ε, αυστηρές πολιτικές λιτότητας. Όχι, είναι το άλλο σκέλος. Είναι ο προπολογισμό που είναι φιλικός προς την οικονομική μεγένθηση. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Τώρα για τις τράπεζες, τα ομόλογα κτλ. Τα δημόσια ομόλογα είναι επικίνδυνα, είναι ένα γεγονός. Δεν ήταν επικίνδυνα μέχρι τις αρχές της κρίσης, τώρα είναι. Ένας καλός επόπτης θα έπρεπε να αναγνωρίζει αυτό το κίνδυνο. Είπαμε όμως και καταλήξαμε στο ότι αυτό πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα ώστε να διατηρήσουμε μια ισότιμη κατάσταση με τις τράπεζες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτές ή δεν έχουν καθόλου κίνδυνο ή πάρα πολύ χαμηλό. Γεγονός είναι ότι αρνούνται κατηγορηματικά να μιλήσουν για στάθμιση ή οποιοδήποτε τρόπο που θα περιόριζε την έκθεσή τους σε δημόσιο, σε δημόσιο ομόλογα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή της Βασιλείας. Αυτή είναι η μία πτυχή. Δεύτερον, θα έπρεπε την πρόοδο αυτή σε αυτό το μέτωπο να την κάνουμε χωρίς να επηρεάζεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι ένα άλλο παράδειγμα. Το είπα και πριν για κάτι άλλο, ότι δεν θέλουμε το φάρμακο να είναι χειρότερο από την ασθένεια. Λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος για τις δυνατές τράπεζες, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν συζητήσαμε για κούρεμα ή ε, ποσοτικούς περιορισμούς, συγκέντρωση κτλ. Όλα αυτά εξετάζονται, αλλά δεν έχει υπάρξει προσανατολισμός προς το παρόν καθόλου. Νομίζω ότι απάντησα σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Φιλίπ Λάμπερτς. Πρόεδρε, μέχρι την παγκόσμια οικονομική κρίση, είχαμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που άφησε το χρέος. Η ποσοτική χαλάρωση και οι πολιτικές αυτές πρώτα από το ΦΕΔ και μετά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βοήθησαν για να σταματήσει αυτός ο εθισμός στο χρέος. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος για το δημόσιο χρέος όσο για εκείνο του ιδιωτικού τομέα, των οικοκυριών, και τα λοιπά. Αναφερθήκατε και στο στεγαστικό κλάδο και άλλα. Λοιπόν, μήπως κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έχουμε αυτό το μοντέλο που μας αρέσει τόσο πολύ, αλλά με τη δημιουργία χρήματος, που είναι πολύ βασικό για τον ιδιωτικό τομέα, τι γίνεται. Με άλλα λόγια, η δημιουργία χρήματος, και εσείς βοηθήσατε βέβαια σε αυτό, η δημιουργία χρήματος εξακολουθεί να είναι προνόμιο του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, μήπως εγώ βλέπω κινδύνους που εσείς δεν βλέπετε, εσείς κανονικά είστε σε καλύτερη θέση για να ξέρετε. Αλλά ειλικρινά, εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου καλά όταν βλέπω αυτά που βλέπω. Πρόεδρος, Ντράγκη, απάντηση. Ας πάμε λίγο πίσω, πριν από την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση δημιουργήθηκε από επεκτατική νομισματική πολιτική που ακολουθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ή μήπω ήταν το αποτέλεσμα μια συστηματικής καταστροφής των κανονισμών που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 και μετά. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο είναι περισσότερο από ότι το πρώτο. Οπότε τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η επεκτατική νομισματική πολιτική ήταν αναγκαία για να έχουμε ανάκαμψη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία και αλλού. Οπότε από αυτή την άποψη το γεγονός ότι τα επιτόκια ήταν χαμηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιούργησε περισσότερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από ότι αν είχαμε μαζικά αποτυχίες και συνεχιζόταν η ανεργία, η ύφεση και ο αποπληθωρισμός. Συνεπώς, αυτή είναι η απάντηση. Όμως, αν πιο συγκεκριμένα δούμε κατά πόσο το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε στην Ευρωζώνη, η απάντηση είναι όχι και τόσο πολύ. σε κάποιες αγορές αναδυόμενες στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείε, ναι, στην Ευρώπη όχι τόσο πολύ. Στην πραγματικότητα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, τα χαμηλά επιτόκια χρησιμεύσαν για να επαναχρηματοδοτήσουν, να αναχρηματοδοτήσουν το υπάρχον χρέος. Συγχρόνως συνέχιζε η ανάπτυξη, οπότε η σχέση χρέους και ανάπτυξης έπεσε σε ένα βαθμό. Τώρα το, το δημόσιο χρέος όχι τόσο. Αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις χώρες, το χρέος στην Ευρωζώνη πέφτει από το 2016 συνολικά. Το ιδιωτικό χρέος μετρίως αλλά μειώνεται. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτή η καθοδική πορεία. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πάντω, τα χαμηλά επιτόκια είναι αναγκαία για να συμμορφωθούμε προ την εντολή μα. Αν υπάρχουν κίνδυνοι σταθερότητα επειδή η, ο ιδιωτικό τομέα έχει κίνητρα να αυξήσει το χρέο του, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μακροπροληπτικά μέτρα. Μα δεν σα ανησυχεί η έκθεση των Ευρωπαίων παικτών εκτός Ευρώπης. Αναφερθήκατε στην Κίνα, ίσως και Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί θυμηθείτε τι έγινε το 2007. Απάντηση, ναι, πράγματι. Υπάρχουν κάποια τμήματα δανεισμού, μόχλευσης ή οι μεγάλες ε, αποδόσεις από το χρέος, αλλά τα προβλήματα αυτά είναι κυρίως στις Ηνωμένε Πολιτείε, όχι τόσο εδώ και εμείς έχουμε μη τραπεζικό τομέα που εκτίθεται στα ίδια προϊόντα. Τα CLOs που τώρα έχουν επανέλθει, ενώ είχαν εξαφανιστεί. Ναι, έχουμε κάποια στοιχεία ανησυχίας από το δεύτερο τμήμα. Ενώ το πρώτο ήταν κάπως καλύτερα. Μιγγέλ Βιέγας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα. Τις... Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Για την Πορτογαλία γίνεται λόγος για εκατοντάδες χιλιάδων ε, δανειακές συμβάσεις που ξεπουλούν οι τράπεζες της Πορτογαλίας σε funds, επενδυτικά ταμεία, και που με βάση και τις πολιτικές της λιτότητας, όταν κάποιος ε, δεν έχει μπορέσει να ξεπληρώσει το δανειό του, βρίσκεται τελικά να πληρώνει ακριβά, πολύ ακριβά την ύφη. Ε, προς τον κύριο Ντράκη λοιπόν η ερώτηση πολύ συγκεκριμένα. Φαίνεται να μεριμνάτε ιδιαίτερος για τις τράπεζες, λιγότερο για τα νοικοκυριά όμως. Και διαρωτώ με, Μήπως ε, με την πώληση αυτών των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων στα φαντς και εκθέτεται υπερβολικά τα νοικοκυριά και ξεπουλάτε φτηνά, πολύ φτηνά αυτά τα ακίνητα και επίσης τα δάνεια υψηλού κινδύνου που βλέπουμε ορισμένες επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν πολύ συχνά. Πώς τα βλέπει η ΕΚΤ. Τα λεγόμενα δάνεια μόχλευσης, leverage loans, ε, φαίνεται και μας το λέει και η Τράπεζα της Αγγλίας ότι είναι σε επίπεδα πάρα πολύ ψηλά, πολύ υψηλότερα και από ό,τι ξέραμε πριν από την κρίση. Δεν σας ανησυχεί αυτό, κύριος Δράγκη. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ με παρεξηγήσετε. Ε, δεν ισχύει ότι μεριμνώ για τράπεζες και όχι για ανθρώπους. Αλλά εάν έχω υψηλό απόθεμα ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων, και το σύστησαμε και νωρίτερα, Πρέπει να κάνω διάκριση μεταξύ αυτού που είναι γνήσια φτωχός, αυτού που πράγματι έχει πληγεί, είναι αδύναμος ε, δανειολήπτης και εκείνου που είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής, που δεν θέλει να πληρώσει. Επομένως πρέπει να φροντίσω τον φτωχό δανειολήπτη, να τον βοηθήσω να ξεπληρώσει την τράπεζα. Άρα με ρημνώ για τον πολίτη, οπωσδήποτε και με ρημνώ για τον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα και γι' αυτό επιπλέον πρέπει να μεριμνήσω να μην καταστρέψω το τραπεζικό μου σύστημα, το τραπεζικό σας σύστημα. Γιατί αν το τραπεζικό σύστημα καταστραφεί δεν θα μπορεί να προσφέρει δάνεια, να δίνει δάνεια, να χορηγεί δάνεια στην οικονομία. Επίσης, τράπεζες με υψηλή μάζα μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως και εκείνες που δεν έχουν, ε, ε, δεν μπορούν μάλλον, αυτές που έχουν υψηλή μάζα ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων, δεν μπορούν να χορηγούν δάνεια ή τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό που μπορούν εκείνε που δεν έχουν με εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, θα τα, θα τα δίνουν με τρόπο πολύ ισχνό, πολύ ψοφοδέη και τελικά που δεν θα υποστηρίζει την οικονομία. Επομένω, ναι, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά διαφορετικό τρόπο τα κοινωνικά προβλήματα χωρί να πληγεί, χωρί να ζημιωθεί το τραπεζικό σύστημα. Αλλά ναι, συμφωνώ, πρέπει να ρυθμιστεί το κοινωνικό ζήτημα. Ευχαριστώ Κύριο Βάλη. Πρόεδρε, κύριος ε, για τη δεύτερη ερώτηση. Μα την έχω απαντήσει και νωρίτερα. Βεβαίως και βεβαίως συμφωνούμε με την Bank of England ότι πρέπει να παρακολουθούμε εκ του και να φροντίζουμε να μην χάνουμε την επαγρύπνηση ως προς τον δανεισμό μόχλευσης και τα συναφή προϊόντα που πολλούνται προκειμένου να ενισχύσουν την απόδοση των επενδύσεων. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να διαγνωστεί γιατί δεν, δεν το προξενεί το τραπεζικό σύστημα, αλλά τα μη τραπεζικά ιδρύματα. Ευχαριστώ Μάρκο Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω και εγώ με την ερώτηση του συναδέλφου Βιέχας για τα μη εξυπηρετουμένα δάνεια, καθώς ε, πρόσφατα, όπως άλλωστε γνωρίζετε, φαντάζομαι, έγιναν, δόθησαν κάποιες ενδείξεις από το, σύστημα, το νέο σύστημα ε, το νέο προληπτικό σύστημα και για την Ιταλία. Ανισχυτικά μηνύματα που δείχνουν ένα συστημικό πρόβλημα βεβαίως εφόσον υπάρχουν τόσο πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι υπήρξαν ε, χώρες οι οποίες μπόρεσαν στο εγγύς με παρελθόν να βρουν λύσεις για να διαχειριστούν το πρόβλημα, ενώ η Ιταλία δεν αξιοποίησε δημόσιους πόρους για να το κλείσει. Διαρωτώ με λοιπόν πώς είναι δυνατόν να συνδυάζεται ένας μηχανισμός τόσο προβληματικός. και να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται η μεγάλη μάζα των μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων αυτό που γίνεται δεν συνιστά υγιή διαχείριση του προβλήματος. Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντική και η υποτίμηση των ε, αξιών των ακινήτων αυτών ε, που προκύπτει λόγω του εις του προβλήματος και βέβαια τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δανειολήπτης. Ερωτώ λοιπόν εάν υπάρχουν ε, εκτιμήσεις σε σχέση με ένα συστημικό πρόβλημα που θα μπορούσε να ε, διατηρηθεί στο χρόνο και να επεκταθεί στο χώρο και αν έχετε σημειώσει σε σχέση και με την πτώση των τιμών των ε, μετοχών κίνδυνο για τις ε, τράπεζες από την έκθεση σε δεύτερου και τρίτου επίπεδου προβλήματα ρευστότητας. Σε σχέση με την επιδείνωση λοιπόν αυτών των ενεργητικών, σκοπεύετε να κάνετε κάποια ανακοίνωση και τι βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ και στις δύο περιπτώσεις νομίζω την ερώτηση πρέπει να απευθύνεται στον μηχανισμό SSM και βεβαίως φαντάζομαι το ο πρόεδρος του θα είναι στη διαθέση σας για να δώσει απαντήσεις στην προσοχή ακρόαση αλλά κάποιες γενικές παρατηρήσεις και για τα δύο αυτά θέματα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρώτον, ε, ναι, πρέπει να δοθούν απαντήσεις, είναι πρόβλημα, στο πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γιατί αποδυναμώνουν τις τράπεζες, μειώνουν το δυναμικό των τραπεζών να χορηγούν δάνεια, αναμφίβολα. Οι τράπεζες που έχουν μάζα μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πιο ασθενείς από αυτές που δεν έχουν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει ε, για το πρόβλημα αυτό η απάντηση που θα δοθεί να είναι τέτοια που να καταστρέψει το τραπεζικό σύστημα. Η απάντηση είναι ουχή. Άρα και πάλι ε, αναζητείται μια λεπτή ισορροπία. Δεν πρέπει το φάρμακο να σκοτώσει τον ασθενή. Δεν θέλουμε το φάρμακο να είναι πιο βαρύ από την αρρώστια. Και άλλωστε και η Επιτροπή σας έχει δραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο Βοήθησε δηλαδή τις πλευρές να καταλήξουν σε μια λογική αλλά και αποτελεσματική επιλογή πολιτικών λύσεων. Σημαντικό όμως είναι και να αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει, πρέπει να επιληθεί. Επίπεδο 2, επίπεδο 3, ε, στοιχεία ενεργητικού δεύτερου και τρίτου επίπεδου. Βεβαίω και είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα, βεβαίω και μα απασχολεί, το συζητούμε. Δεν προβλέπουμε αυτή τη στιγμή ανακοίνωση στο βαθμό που εγώ μπορώ να το γνωρίζω. Πρέπει εδώ να είμαι προσεκτικός στο πώς θα το πω, γιατί μπορεί ο SSM να σκέφτεται να κάνει ανακοινωθέν, αλλά εγώ ενημέρωση τέτοια δεν έχω. Σας ευχαριστώ που μνημονεύσατε άλλωστε και, το, και την παρούσα επιτροπή και τον ρόλο της. Ο κύριος Γκέρολτ, κύριε Πρόεδρε, ερώτηση για την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων και ήδη κάπως θίξατε το θέμα. Οι τιμέ των ακινήτων ήταν πάντοτε πηγή ανησυχία σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των συστημικών κινδύνων και στην ε, η κρίση των subprimes ήταν επειδή έσκασε η φούσκα στην αγορά στέγης στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από το φτηνό χρήμα που διέθεσε η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών στην αγορά. Στην έκθεσή σας προμηνός αναφέρεστε στις τιμές ακινήτων στέγης σε πολλές χώρες μέλη φαίνεται να είναι υπερτιμημένες. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα συσχετισμός ανάμεσα στην πολιτική επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όλοι συμφωνούμε ότι μια παρόμοια φούσκα στην αγορά ακινήτων όπως τότε στις ΗΠΑ αποτελεί συστημικό κίνδυνο. Δύο ερωτήσεις. Πόσο πολύ, πολύ μπορεί να αυξηθεί η ε, τιμή των ακινήτων μέχρι ότου θεωρήσετε ότι είναι συστημικός κίνδυνος και δεύτερο το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου προβαίνει σε αξιολόγηση και θεωρεί ότι είναι αρκετά επικίνδυνη η κατάσταση ώστε να χρησιμοποιήσει εργαλεία και ποια θα ήταν αυτά. απάντηση του κ. Ντράγκη. Ε, δεν συμφωνώ με την εκτιμήσή σας ότι το φτηνό χρήμα της ΦΕΔ αποτέλεσε την αιτία για την δημοσιονομική κρίση στις ΗΠΑ. Δεν θα σας ευνηδιάσει επομένω αν σας πω ότι δεν θεωρώ ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αλλάξουν διότι είναι υπερτιμημένη η αγορά κινήτων. Δεν θα ήταν το σωστό μέτρο για να ληφθεί αυτό. Όταν υπάρχει υπερτίμηση μιας συγκεκριμένης αγοράς η αγορά κινήτων κατοικίας είναι υπερτιμμένη μόνο σε ορισμένες μεγάλες πόλεις και σε ορισμένα τμήματα της Ευρωζώνης. Παρόλο που βλέπουμε ότι αυξάνονται περισσότερο τιμές ακινήτων από ό,τι στο παρελθόν. Δεν βλέπουμε αυξημένη, ε, αυξημένο δανεισμό. Όταν βλέπουμε αυξημένο δανεισμό, βλέπουμε ότι εν μέρη είναι για την ε, αγορά ακινήτων. Πιο πολύ βλέπουμε όμως τα εμπορικά ακίνητα να ε, είναι υπερτιμμένα. Πάντως, ξαναλέω, για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά χρειάζεται μακροπροληπτική πολιτική, όχι νομισματική πολιτική. Να κάνει κανείς κάτι άλλο θα σήμαινε ε, να αντιταχθεί στην εντολή μας να χρησιμοποιεί δηλαδή νομισματική πολιτική για να εξασφαλίσει την νομισματική σταθερότητα, ότι υπάρχουν οι όροι για να ε, είναι ο πληθωρισμός αυτός τον οποίο στοχεύουμε, για να λύσετε ένα πρόβλημα σε ένα τομέα χρησιμοποιείται μακροπροληπτική πολιτική και αυτό το εξετάζει το Συμβούλιο Στατιστική Συστημικού Κινδύνου Ευχαριστώ κύριε Μπερέση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπό την ιδιότητά σας προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων θέλω την εκτίμησή σας για την εντολή που έδωσε η Επιτροπή μας για την αναθεώρηση της διακυβέρνησης του οργάνου αυτού. Η δικιά μου γνωμοδότηση, όπως ξέρετε, δεν προχώρησε πολύ, αλλά θέλω τη δικιά σας εκτίμηση. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε με μία αξιολόγηση των ε, έργων ε, της αρχής, των επιπτώσεων της πολιτικής που ασκεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων και στις ανταλλαγές που είχαμε και με τον κύριο Ντελαροζιέρ, ε, καταλάβαμε ότι ουσιαστικά θα έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί οι μελέτες του οργάνου αυτού δεν θα πρέπει να μείνουν ακαδημαϊκά χαρτιά σε ένα σιρτάρι, αλλά θα έπρεπε να δίνεται και κάποια συνέχεια, να λαμβάνονται υπόψη οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι. Οπότε πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη της χρηστής διακυβέρνησης. Έχει γίνει καλή χρήση της ευκαιρίας αυτής. Δεύτερον, θέλω να φερθώ σε κάτι που θίξατε λίγο, και είναι η ε, κίνδυνοι που εντοπίσατε και αναπτύξατε. Μάλιστα στην προηγούμενη ανταλλαγή που είχαμε μεταξύ μας, πρόκειται για το κίνδυνο της εμπορικής στέγασης. Και τώρα αναφερθήκατε και πάλι σε αυτό πριν από λίγο. Εγώ θέλω να ξέρω τι συστάσεις συγκεκριμένα έχετε εσείς σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία ε, θα πρέπει να ασχοληθούν ε, οι G7, οι G20. Γιατί δημιουργήσατε ανησυχία έτσι όπως εκφραστήκατε για το τι κάνει ο στεγαστικός ο κλάδος και τι κινδυνεύει να κάνει στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μπορείτε να είσαστε πιο συγκεκριμένους λοιπόν για το πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την παγίδα. Για την πρώτη ερώτηση. Η όλη συζήτηση ξεκίνησε με την αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δεν υπογράμμιζε τους κινδύνους από τα χαμηλά επιτόκια όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα. Και το συμπέρασμα ήταν ότι προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων, η διακυβέρνηση θα έπρεπε να αλλάξει. Δεν είναι αλήθεια γιατί ναι, το Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων είπε ότι από τα χαμηλά επιτόκια, μάλλον ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τα χαμηλά επιτόκια. Επίσης δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων, γιατί το δεύτερο όργανο είναι μείον 2 από τους 36. Οπότε θα έλεγα ότι η διάγνωση ήταν λανθασμένη. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ο συλλογισμός δεν ήταν σωστός. Οι συνέπειες, ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, θα ήταν η αλλαγή στη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνου, θα καταστούσε το όργανο αυτό πιο αδύναμο στο να φέρει σε πέρα στην εντολή του και όχι περισσότερο ικανό να φέρει σε πέρα στην ε, εντολή του. Η φωνή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων, εφόσον είχαμε ακολουθήσει κάποιες από τις προτάσεις που είδα, τότε θα επικρατούσε περισσότερη σύγχυση. Γιατί αν έχετε πολλές και πολλαπλές φωνές που μιλούν για την οικονομική σταθερότητα και τα ζητήματα ε, προληπτικής πολιτικής, θα ήταν πιο δύσκολη κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων πάντως είναι στη διάθεσή σας να ακολουθήσει τις προτάσεις σας και να φέρει σε πέρα στο έργο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είμαστε ανοιχτοί για να υπάρξει βελτίωση σε όλους τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Αλλά για να απαντήσω συγκεκριμένα για την αλλαγή στη διακυβέρνηση, αυτή δεν θα ήταν η σωστή απάντηση. Τώρα για τον κίνδυνο όσον αφορά την ε, εμπορική στέγαση. Εδώ το στοιχείο κλειδί είναι ότι οι κίνδυνοι αυτοί, ναι, αυξήθηκαν, αλλά ο βασικός παράγοντας δεν είναι το τραπεζικό σύστημα, είναι το μη τραπεζικό. Και η θέση του Συμβουλίου Συντημικών Κινδύνων που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επέκταση του πεδίου εφαρμογής της μακροπροληπτικής ε, πολιτικής και στον μη τραπεζικό τομέα παραμένει πρέπει να επεκτείνουμε και την ομοθεσία για να συμπεριλάβουμε και άλλους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και παράγοντες πέρα από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και στην περίμετρο, για να λυθούν υπόψη στην μακροπροληπτική πολιτική. Και προς το παρόν έχουν εντοπιστεί αυτοί οι κίνδυνοι και δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να δράσουμε σε αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Ολοκληρώνουμε έτσι και αυτό το δεύτερο τμήμα της συνάντησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον τόσο ενδιαφέροντα νομισματικό διάλογο και το διάλογο με το Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων. Σας ευχαριστούμε ξανά για τη συνεργασία σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ.